Dear colleagues. Συνάδελφοι και συναδελφέ, ας μην περιμένουμε άλλο. Ξέρω ότι έρχεται, έρχεται ακόμα κόσμος, αλλά δεν μπορούμε να απεργηθυστερήσουμε περισσότερο. Σας καλωσορίζω σε αυτήν την κοινή συνεδρίαση της ΠΕΡΙΦ με την ΚΟΤΕΡ της Επιτροπής Περιφερειών. Γι' αυτό έχω και τον διπλανό μου εδώ. Είναι ο συμπρόεδρος ο κύριος Μάρικ Βόσνιακ. Αποφασίσαμε φέτος την κοινή μας συνεδρίαση να, στην κοινή μας συνεδρίαση να θίξουμε τέσσερα κύρια θέματα του βασικού πλαισίου για την πολιτική συνοχή δηλαδή πρώτον η πολυεπίπεδη governance καθώς και ο δεοντολογικός κώδικς. Μετά θεματική συγκέντρωση τρίτον περιφερειακή διάσταση και τέταρτον το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που είναι αυτό το καινούριο εργαλείο που έχουμε για καλύτερο συντονισμό στο μέλλον. Δεν χρειάζεται, αλλά ας το ξαναπώ, ότι συνεδριάζουμε σε μια κρίσιμη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ήδη έχουμε ήδη διαπραγματεύσεις ως συνομοθέτες για το νέο ρυθμίστικο πλαίσιο και επίσης ως κοινοβούλιο γνωμοδοτούμε και μπορούμε να ασκήσουμε και βέτο στις διαπραγματεύσεις των πολιετών δημοσιονομικών πλαισίων. Οι δύο διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή θα είναι αποφασιστικές για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Εμείς ως Κοινοβούλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχουμε το δικαίωμα να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνε, Δηλαδή νομοθετούμε υπό τη λεγόμενη κανονική διαδικασία, δηλαδή για όλους τους κανονισμούς για την Ευρωπαϊκή Συνοχή, είναι συνομοθέτης το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο. Οι διαπραγματεύσεις είναι πραγματικά διαπραγματεύσεις λοιπόν και γι' αυτό πρέπει να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς που να μην ε, ε, αποδυναμώνουν αυτή την πολιτική. Για μας είναι σημαντικό. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, είμαστε στεναρός υπέρ των εταιρικών δεσμών και σχέσεων partnership δηλαδή. Όχι μόνο ως προς τη δημοκρατική νομιμότητα της πολιτικής αυτής, αλλά και για να είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι επαρκής. Επίσης υποστηρίζουμε την ευελιξία που θα ε, επέτρεπε τη μετάφραση των στόχων της Ευρώπης του 2020 σε, σε επενδυτικά προγράμματα που να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες πόλεων, τοπικών κοινοτήτων, περιφερειών, ευελιξία λοιπόν η οποία να λύνει περισσότερο καλύτερα τα προβλήματα. Και ελπίζω ότι όλοι εδώ μέσα είναι υπέρ του λεγόμενου better spending θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται και για καλύτερη επένδυση, όχι μόνο για καλύτερη δαπάνηση. Σύντομα λοιπόν για αυτά τα τέσσερα θέματα θα συζητήσουμε σήμερα. Για την ε, δε πολυεπίπεδη governance θα ήθελα να πω ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την έννοια της ε, συνεργασίας δεν είναι κάτι καινούριο βέβαια. Η εταιρική σχέση και η συνεργασία υπήρχε και πριν. Υπάρχουν ακόμη ελλείψεις στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής αυτής αρχής και θα θέλαμε στον κανονισμό να υπάρχουν και ορισμένες ρήτρες ασφαλείας για να προστατευτούμε για να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Επίσης, θα θέλαμε στον κανονισμό να δίνεται περισσότερος ρόλος στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να υπάρχει μια εταιρική συμφωνία έτσι τη λέμε εμείς όχι συμβόλαιο αλλά συμφωνία που να μας επιτρέπει να συνδεόμεθα με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων. Επίσης θα θέλαμε πιο καλά καθορισμένο κατάλογο των εταίρων. Για ναι, το δεύτερο θέμα θεματική συγκέντρωση θα ήθελα να πω ότι από την αρχή, από την αρχή εδώ στο Κοινοβούλιο πάντα ήμασταν υπέρ της, ε, του συνδυασμού με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 για να συνεισφέρουν όλα αυτά με αυτό τρόπο στο, στην επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όμως και αλλά τα καταλαβαίνουμε ταυτόχρονα ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο αν υπάρχει αρκετή ευελιξία που να δίνει στις περιφέρειες και τους δήμους και κοινότητες περισσότερες δυνατότητες για να μπορούν να προσαρμόσουν τα προγράμματα στις ιδιαιτερότητες των. Αυτό το τονίζουμε πάντοτε. Τρίτον, η περιφερειακή διάσταση εδώ προτείνουμε επίσης πολλές αλλαγές στον κανονισμό για να ενισχυθεί η περιφερειακή αυτή διάσταση στην δομή, στο μηχανισμό Παράδειγμα, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σύνδεση μεταξύ αστικών και υπεθρίων περιοχών και τα νέα όργανα για καλύτερο συντονισμό των προγραμμάτων με συνδυασμό με τα μακροοικονομικά συμφέροντα και των περιφερειών και τοπικών κοινοτήτων. Θέλουμε δηλαδή πιο ορατή και χρηματικά περιφερειακή συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θέλουμε για πρώτη φορά έχουμε για πρώτη φορά τις κοινέ διατάξεις και κανόνες που διασφαλίζουν τη συνέπεια και ακριβώς τη συνοχή μεταξύ και των πέντε ταμείων που έχουμε στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Και για να υπάρξει αυτή η καλύτερη συνεργασία και συνέργεια πρέπει να ξέρουμε πώς μπορούμε καλύτερα να συνδυάσουμε και τα πέντε τα μία. Αυτή είναι η δική μου εισήγηση και τώρα θα δώσω το λόγο στον συμπρόεδρο, στον πρόεδρο της Επιτροπής Κοτέρ, Μάρικ Βόσνιακ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ και συμπροεδρεύω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 ten Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να συναντηθούμε εδώ με όλους όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική συνοχής. Και η στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πολύ κρίσιμη, διότι έχουμε τις ε, συζητήσεις ε, για τον προϋπολογισμό, μεταξύ άλλων. Βέβαια, ο προπολογισμό, όπω καταλαβαίνετε, θα επηρεάσει τα μάλα και το μέλλον τη πολιτική συνοχή. Αν δεν είναι ο σωστό, αν δεν είναι καλό αυτό ο προπολογισμό, τότε όλοι οι κανόνε που μα αφορούν θα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής θα πρέπει να διορθωθεί και ε, γι' αυτό το λόγο εμείς ε, Συζητάμε με την Επιτροπή των Περιφερειών, ε, συμμετέχουν όλοι από κοινού, γιατί είναι πεπισμένοι ότι η πολιτική συνοχής ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και θέλουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτική συνοχής. Αυτό, μεταξύ άλλων, ε, εκφράζεται με την στρατηγική Ευρώπη 2020. Η Επιτροπή των ε, Περιφερειών ε, κατέθεσε την άποψή της και εντωμεταξύ προετοιμάζουμε μία έκθεση για για το κοινό πλαίσιο. Εγώ έχω την τιμή σε αυτόν τον τομέα να είμαι βασικός εισηγητής και ελπίζω ότι η γνωμοδότησή μας θα εγκριθεί από την Επιτροπή των Περιφερειών κατά τη διάρκεια της ε, Ολομέλειας του Νοεμβρίου. Ε, γνωρίζουμε ότι οι μέχρι τώρα γνωμοδοτήσεις ε, πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε όλες τις απόψεις. Επίσης όλα τα θέματα τα οποία μέχρι τώρα δεν εκφράζονται στις ε, διάφορες προτάσεις. Όλα αυτά τα σχέδια θα τα ανασυντάξουμε και στις αρχές του έτους, ε, τον Ιανουάριο, ε, θα καταθέσουμε και εμείς τη νέα μας γνωμοδότηση για την πολιτική συνοχής και θα τα υποβάλουμε στο Συμβούλιο. Εγώ ε, προετοίμασα μαζί με τους συναδέλφους μου ε, τις απόψεις μας για τη σημερινή συνάντηση. Ε, έχουμε αναλύσει τις απόψεις του Κοινοβουλίου και όλα αυτά τα έχουμε συνοψίσει σε ένα κατάλογο 11 σελίδων. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στη θέση να μπορώ να διαπιστώσω ότι όλα αυτά τα θέματα εκφράζουν τις απόψεις μας, συμπίπτουν με τις απόψεις μας. Ελάχιστες είναι οι διαφορές. Νομίζω όμως ότι παρόλα αυτά ε, μπορούμε να υποφεληθούμε από το ότι έχουμε ένα τόσο ισχυρό εταίρο, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατόπιν τούτου είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε τις απόψεις μας ε, να τις ε, εκφράσουμε άμεσα είτε στους εισηγητές είτε στον πρόεδρο, στην πρόεδρο της Επιτροπής. Χαίρομαι που έχετε τίνει ευήκονους προς εμάς, διότι σας είπα ότι επιθυμούμε να έχουμε έναν ισχυρό εταίρο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ας δούμε λιγάκι τι θέλω να σας επισημάνω. Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι αυτονόητο ότι η πολιτική συνοχής για μας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Στην Επιτροπή των Περιφερειών δεν άκουσα κάποιος ε, να επιθυμεί να περιοριστούν οι δαπάνες στο μέλλον. Και αυτό οφείλεται στο ότι όλες οι επιτροπές έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν περαιτέρω. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ε, υποστηρίζουμε τις ε, περιφέρειες εκείνες οι οποίες βρίσκονται σε μεταβατική φάση, οι οποίες ε, αναπτύχθηκαν περαιτέρω τα τελευταία χρόνια και όπου το κατακεφαλή ΑΕΠ είναι κατά τη ψηλότερο, δηλαδή από 75 μέχρι 90%. Όμως πρέπει να σας πω ότι γνωρίζουμε επίσης ότι οι περιφέρειες αυτές πρέπει να στηριχτούν περαιτέρω γιατί επουδενή δεν μπορεί να ισχύει η επιτυχία που έχει σημειωθεί να οδηγήσει στην ε, μείωση της υποστήριξης απέναντι σε αυτές τις ε, περιφέρειες. Αυτό που επίσης ε, έχει σημασία και είναι, θα έλεγα μάλιστα, παράδοση στην Επιτροπή των Περιφερειών, το λοιπόν που έχει σημασία είναι να ε, ταχθούμε πέρ μιας ε, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά διάρκεια των ε, επιτροπών της ΚΟΤΕΡ, εμείς εγκρίναμε έναν κώδικα συμπεριφοράς και αυτόν τον κώδικα θα τον παρουσιάσουμε κατά τη διάρκεια τη επόμενη συνεδρία τη Επιτροπή των Περιφερειών. Θα ψηφίσουμε από αυτού και νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταστεί σαφέ ότι η δική μας άποψη, η γνώμη της Επιτροπής των ε, Περιφερειών πρέπει να εισακούεται καθ' όλη τη διάρκεια της ε, νομοθετικής διαδικασίας. Εξίσου σημαντικό είναι για μας να στηρίξουμε και την στρατική Ευρώπη 2020. Γνωρίζουμε ότι στις ε, διαπραγματεύσεις αυτό που είναι σημαντικό είναι ε, να ασχοληθούμε με την ε, εκταμείευση και την κατανομή των κονδυλίων. Προφανώς εδώ είναι απαραίτητο να υπάρχει συμβιβασμός. Κατά τα άλλα, οφείλουμε να έχουμε και την απαραίτητη ευελιξία κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Εγώ προσωπικά ε, ηγούμε, είμαι επικεφαλής σε, μια κάποια ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, απαιτήσει του μέλλοντος. Τα προγράμματα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα ε, στις ε, δικές μας τις αποτήσεις, απαιτήσεις ε, και στις συνθήκες, γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε μέσα σε αρτηριοσκληρώσεις και αγκυλώσεις. Η τοποθέτηση της Επιτροπής των Περιφερειών είναι σαφέστατη κυρίως όσον αφορά στις, ε, στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Κυρίως στην ε, διασύνδεση της ε, συνοχής με τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Φοβούμαστε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ ή αν υπάρξει πολύ στενή διασύνδεση με το μακροοικονομικό περιβάλλον, τότε εκείνοι που εφαρμόζουν τα προγράμματα, δηλαδή εμείς οι περιφέρειες, δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξελιχθούν περαιτέρω όπως το επιθυμούν. Η πολύ στενή διασύνδεση, κατά την άποψή μας, δεν είναι επωφελής. Εξάλλου προσβλέπουμε σε μια κάποια ε, σταθερότητα της ε, διαδικασίας ε, προγραμματισμού. Ελπίζουμε κυρίως ότι η οικονομική κατάσταση θα ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων. Κυρίως ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αν έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, στα προγράμματα, αυτό θα αποτελεί για μας ε, εμπόδιο. Δεν υπάρχει ασφάλεια σχεδιασμού και κατόπιν τούτου είναι πολύ δύσκολο ε, λόγω αυτής της ε, ασταθούς ε, κατάστασης να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε με επιτυχία. Εξάλλου τα σώμεθα κατά ενός συστήματος επιβράβευσης για την δημιουργία αποθεμάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι το σύστημα μπορεί να οδηγήσει ε, στο να αναδιαμορφωθούν οι στόχοι. Δηλαδή οι στόχοι γίνονται πιο περιορισμένοι για να δημιουργηθεί ένα απόθεμα. Και αυτό δεν νομίζουμε ότι είναι σωστό. Τέλος, όσον αφορά την απλούστευση ε, από το πρίσμα μιας ε, οργάνωσης η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή των προγραμμάτων, πρέπει να πω ότι αναμφίβολα είναι πολύ σημαντικό να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Επ' αυτού γίνεται πολύ συχνά λόγος, όμως δυστυχώς οι διαδικασίες γίνονται όλο και πιο δύσκολες, όλο και πιο περίπλοκες, διότι ξεκινάει κανείς από την παραδοχή ότι με περίπλοκες ρυθμίσεις αποκλείονται οι κακές πρακτικές. Όμως αν υπάρχει ακριβής διατύπωση των διαδικασιών, ακόμα και αν υπάρχει ακριβής διατύπωση, ε, παρόλα αυτά η εφαρμογή ενδέχεται να είναι δυσκολότερη. Ή θα μπορούσα να το πω αλλιώ. Ναι, πράγματι πρέπει να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες Αυτός είναι κατ' ουσίαν ο μοναδικός στόχος που πρέπει να έχουμε κατά νου και νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα ελπιδοφόρος. Σήμερα εκπροσωπούνται εδώ και οι συγητές των διαφόρων τομέων πολιτικής συνοχής. Ε, αυτοί είναι στη διάθεσή σας. Ευχαρίστω να απαντήσουν στις ε, ερωτήσεις σας ε, και ευχαρίστω να ανταλλάξουμε απόψεις. Αυτά είχα να πω εν είδη εισαγωγής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώ επειδή έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο, τώρα αρχίζουμε τον αγώνα. Πρέπει να προλάβουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τη σειρά, με τα τέσσερα αυτά θέματα, 15 το πολύ λεπτά για το καθένα. Πρώτο θέμα λοιπόν είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και ο κώδικας εντολογίας. Να ακούσουμε πρώτα από εσά κάποια πράγματα και μετά να ακούσουμε και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε περίπτωση που έχουν να πούν κάτι ή τα μέλη από την Επιτροπή Κοτέρ, ελπίζοντα κυρίως βέβαια από τους εξωτερικούς μας προσκεκλημένους ε, ότι θα θελήσουν να λάβουν το λόγο. Όσοι θέλουν λοιπόν να καταθέσουν μια ερώτηση, παρακαλώ να μην υπερμούν το ένα λεπτό. και ταυτόχρονα να συστηθούν, να μας πούν ποιοι είναι, από πού προέρχονται κτλ. Ξεκινάμε λοιπόν από την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση τη συμπράξη των κώδικα διοντολογία. Υπάρχει κάποιο που θα ήθελε το λόγο να θέσει κάποιο ερώτημα. Uh, we see a European parliamentarian, Ο κύριος Νίλσεν, από ό,τι βλέπω, θέλει το λόγο. Γεν Νίλσεν. Ήμουν 10 χρόνια στην Επιτροπή Κότερη της Επιτροπής των Περιφερειών και ένα θέμα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή των Περιφερειών αλλά και για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η αρχή των συμπράξεων, των εταιρικών σχέσεων. Όπως προτείνεται και όπως ορίζεται είναι αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλή, αλλά εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την έννοια. Πολλέ κυβερνήσει βέβαια δεν συμφωνούν με την αρχή αυτή, γιατί φυσικά έχει να κάνει με αποκέντρωση των εξουσιών. Ως Ευρωβουλευτή πλέον λοιπόν έχω το εξή ερώτημα. Η Επιτροπή των Περιφερειών πόσο δραστήρια κινείται και πώ και αν μπορεί να ασκήσει πιέσει στις κυβερνήσει ώστε να καταλάβουν ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης είναι απολύτως σημαντική για να υλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές. Η Πρόεδρος, παρακαλώ να ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν το θέμα αυτό, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Εσείς παρακαλώ. Σεμπαστέν Κανιέ λέγομαι και εκπροσωπώ Ολλανδικούς ε, φορείς κοινωνικής στέγασης. Μήπω ε, χρησιμοποιούν για την έρευνα και την ανάπτυξη για κυροσκοπικού οργανισμούς αυτά τα κονδύλια. Βλέπω ότι ε, στη χώρα μου υπάρχει ακριβώ αυτή η πίεση να πάνε σε συγκεκριμένου, συγκεκριμένους κορυφαίους ε, οικονομικούς τομείς αυτά τα χρήματα. Πώς για την νομοθεσία ότι υπάρχει μια εξισορρόπηση των εμπορικών συμφερόντων με την ανάγκη να υπάρχουν και μη κερδοσκοπικέ δραστηριότητε, όπω είναι κοινωνική κατοικία, κοινωνικό επιχειρήν, και ποιο θα έπρεπε να είναι εδώ ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα αξιολογεί αυτέ τι συμπράξει σε δημοσιο τομέα. Ευχαριστώ. Any other question? Υπάρχουν άλλε ερωτήσει ή σχόλια για αυτό το θέμα. Ο κύριος Βλάσακ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, θα εκμεταλλευτώ και εγώ τη διερμηνή και θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να ρωτήσω ε, κατά πόσον οι περιφέρειες είναι προετοιμασμένες για το ανώτερο ή ανώτατο επίπεδο συνεργασίας. Στο πλαίσιο της ε, τριμερού συνάντησης ε, εξετάζουμε το θέμα των συμβάσεων παραχώρησης και αυτό σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης ε, θα συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις ε, μαζί με την κυβέρνηση. Έχετε λοιπόν προετοιμαστεί έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις αυτές να είναι ταχύτατες και αποτελεσματικές. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια παρακαλώ. Ερώτηση καμία. Άντε, μια τελευταία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Άκουγα αυτή τη συζήτηση και άκουσα να γίνεται λόγος για partnerships, για εταιρικές σχέσεις, πράξεις, αλλά εγώ θεωρώ ότι τρία είναι τα επίπεδα, το περιφερειακό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε σε δύσκολους καιρούς. Δοκιμάζεται ο κόσμος. Σε αυτά τα τρία επίπεδα, το τοπικό, το περιφερειακό αφενός το εθνικό αφετέρου και τρίτον το ευρωπαϊκό, πολλές φορές χρησιμοποιούνται κάποια προσχήματα για να αποφευθεί η αποκέντρωση. Και μάλιστα για μεγαλύτερη συγκέντρωση των επιπέδων αυτών. Πώς λοιπόν σε αυτή την εταιρική σχέση και σε αυτές τις συνομιλίες σχετικές, πώς μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερο τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ώστε όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο να περιοριστούν. Ξέρουμε βέβαια ότι ορισμένα project εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Πολύ συχνά όμως παραλείπονται από αυτές τις συζητήσεις. Κύριο Σόσφαλτ. Να μιλήσω και εγώ τσέχικα, όπως ο κύριος Βλάσακ ή να μιλήσω αγγλικά. Όχι, θα μιλήσω τσέχικα. Ετέθη το ερώτημα κατά πόσον εμείς ως Δήμοι και κοινότητες είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε εταιρική σχέση. Αν θυμάμαι καλά, η προετοιμασία αυτής της ε, περίοδου, της προγραμματικής περίοδου, βασίστηκε στη συμπερίληψη των ε, δήμων και κοινοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά συνήθως συμβαίνει το, εξή, το εξής. Ε, μας διαβάζονται κάποια έγγραφα και η απάντηση κατ' ουσίαν δίδεται αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη. Και τώρα δεν ομιλώ μόνο εκ μέρου της ε, Τσεχίας. Μας ενδιαφέρει όλους μας ε, να τύχουν επεξεργασίας οι προτεραιότητες, ε, κυρίως εκείνες τις οποίες χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν το λιγάκι τα αναπτυξιακά προγράμματα στην Τσεχία, δηλαδή τα προγράμματα τα οποία έχουν υπόψη τους οι δήμοι και οι κοινότητες, διαπιστώνουμε ότι κατά 40% γίνεται χρήση κοινοτικών κοντιλίων. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει οι αρμόδιες ομάδες να είναι προετοιμασμένες, όπως είπε ο κύριος Βλάσακ, γιατί αλλιώς είναι σαν να εκχωρούμε αρμοδιότητες ως τοπική αυτοδιοίκηση, σαν να πεμπολούμε μάλλον αρμοδιότητες. Όσον αφορά τώρα τη συμπερίληψη σε διάφορα επίπεδα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία ε, λεπτομερής μέθοδος για τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα. Αυτό το λέω εδώ και καιρό. Εγώ τάσομαι υπέρ του να ζητείτε από όλα τα κράτη-μέλη να ορίζουν με ακρίβεια κάθε κεφάλαιο ε, να ορίζουν το τι ακριβώς είναι η εθνική, το εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ορίσουμε καλύτερα τις ε, εκάστοτε ανάγκες, τις οικίες ανάγκες. αντιπρόεδρος της περιοχής Ρον Αλπ στη Γαλλία. Δύο παρατηρήσεις. Πολλά υπόθηκαν, εγώ θα ήθελα να επιμείνω προς τους συναδέλφους ευρωβουλευτές για το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος. Διότι συχνά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Καλό είναι να συμμετέχουν άπαντες και ξέρετε για την διαχείριση και την προετοιμασία των Ευρωπαϊκών Τέμων θα αλλάξουν οι κανονισμοί. Χρειάζεται χρόνος. Και νομίζω ότι θέλετε κι εσείς να υπάρχει χρόνος για αυτές τις ε, συμπράξεις και για τα εθνικά σχέδια δράσης. Εγώ στην περιφέρεια μήτε από σήμερα, το δεύτερο εξάμεινο του 2012, αρχίζω να ε, προσπαθώ να συμμετέχουν οι τοπικοί φορείς. 6 εκατομμύρια κάτοικοι όμως είναι, με πολλούς δήμους, πολλά διαμερίσματα. Χρειάζεται χρόνος, αλλά είναι αποφασιστική σημασία στο χρονοδιάγραμμα. πρέπει να υπάρξουν αυτές οι εθνικές συμφωνίες, πρέπει οι περιφέρειες και η τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετέχουν από την αρχή και να έχουμε και κάποιο χρόνο πριν τον καθορισμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αλλιώς τελικά θα επικρατήσει μια τεχνοκρατική λογική και δεν θα μπορέσει καθόλου να συμμετάσχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Λυπούμε για τον έχω χρόνο γιατί θα ήθελα να πω πολλά άλλα. Επιμένω όμω σε αυτό το θέμα του χρονοδιαγράμματο γιατί αποτελεί προπόθεση για μια πραγματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Γιάνν Όλμπριχτ και ίσως κάποιος άλλος από την Επιτροπή Κότερ και μετά αν όχι θα περάσουμε στα άλλα θέματα. Γιάν, θα ήταν καλό εκτός από την ερώτηση να μας παρουσιάσει λίγο και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωραία, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να θυμόμαστε ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε την όλη φιλοσοφία των ταμείων. Δεν πρόκειται για διαβουλεύσεις, πρόκειται για εταιρικές σχέσεις. δεν θα υπάρχουν εθνικά σχέδια. Στρέφαμε στον προλαλήσαντα. Μόνο η λεγόμενη σύμβαση εταιρική σχέση θα υπάρχει. Partnership contract. Τι σημαίνει αυτό, ποια είναι η φιλοσοφία. Όλοι οι εταίροι συνεργάζονται από κοινού και εκπονούν το έγγραφο το οποίο θα αποτελέσει το πλαίσιο για το όλο σύστημα. Για 7 έτη. Ξέρετε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα όλα αυτά γιατί θα υπάρχουν πολλοί εταίροι. Αλλά αυτό είναι ο μόνο τρόπο δεν είναι ότι έχουμε ένα έγγραφο που εκπονείται από την κυβέρνηση και έπειτα ακολουθεί διαβούλευση. Όχι. Από κοινού όλοι οι εταίροι εκπονούν το έγγραφο. Και όχι μόνο το εκπονούν, αλλά το έγγραφο, το οποίο μπορεί και να τροποποιηθεί σε αυτή την επταετία μέσα, πάλι πρέπει να τροποποιηθεί από όλου του εταίρου. Η αρχή τη εταιρική σχέση σημαίνει, αν διαβάσει κανεί το σχέδιο κανονισμού, που εμεί είμαστε υπέρ εδώ στο Κοινοβούλιο, το είπε και στην αρχή, Όλοι οι εταίροι, λέει, πρέπει να λαμβάνουν μέρος στη διαχείριση κάθε φάσης της διαδικασίας προγραμματισμού και υλοποίησης. Μεγάλη πρόκληση. Πώς όλοι οι εταίροι μπορούν να είναι ενεργοί δραστήριοι και να συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κομισιόν προτείνει αυτόν τον κώδικα διοντολογία, Code of Conduct, και τα κράτη-μέλη πάλι καθόλου τυχαίο δεν είναι που δεν το δέχονται αυτό. Το Συμβούλιο δεν θέλει να υπάρχει ένα σύστημα για όλη την Ευρώπη, ένα κώδικα διοντολογία για όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι σημαντικό. Και υπάρχει και το θέμα των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η Κομισιόν σήμερα θέλει να υπάρχουν αυτές οι συμβάσεις ή συμφωνίες εταιρικής σχέσης μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα, αυτά να γίνουν ταυτόχρονα δηλαδή για να ε, κερδιθεί χρόνος. Εμείς όμως τι προτείνουμε, να γίνουν σε δύο χρόνους αυτά, αλλά βέβαια το στόμα το πρώτα να έχουμε τη σύμβαση αυτή, το συμβόλαιο τέτοια σχέση, να συμφωνηθεί το σύστημα, το σχήμα και μετά να έχουμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Γιατί αν η σύμβαση της εταιρικής σχέσης δεν συμφωνηθεί και δεν εγκριθεί από την Κομισιό, τι θα γίνει μετά με τα επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτά είναι τα ζητήματα είναι εισαγωγή για τα επιχειρησιακά προγράμματα. Είναι το πρώτο τμήμα του πακέτου. Η Κομισιόν θέλει να είναι τμήμα του πακέτου. Εμείς θέλουμε να είναι το πρώτο βήμα, το πρώτο στάδιο. Και εδώ υπάρχει μια ε, διαφωνία. Ο συνάδελφος Βλάσεκ τα είπε πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα και λοιπόν που το λέω. Υπήρξα δήμαρχος ε, ε, και νομάρχης Θέλουμε εταιρική σχέση μεταξύ τοπικού και περιφερειακού. Είναι πρόκληση αυτό. Πρόκληση και για την Επιτροπή των Περιφερειών. Διότι όλο και μεγαλύτερη συζήτηση γίνεται μεταξύ περιφερειών και πόλεων. Όταν η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ρέγγιο, ξέρετε, άλλαξε το όνομα ε, που είχε, γιατί πλέον είναι πολιτική η διεύθυνση αρμόδια για την περιφερειακή αλλά και την αστική ανάπτυξη. Τονίζω πρέπει να υπάρξει μια πραγματική εταιρική σχέση, όχι μόνο μεταξύ κυβερνήσεων και λοιπόν, αλλά μεταξύ όλων μεταξύ τους. Από την πλευρά της Επιτροπής ε, των Περιφερειών, Μιχαλ Σνάιντερ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω κάτι επ' αυτού. Πρόκειται για ένα περίπλοκο και δύσκολο θέμα αυτό που εφήγει. και θα μπορούσε κανείς ε, να κάνει μια ολόκληρη διάληξη για αυτό το θέμα. Κύριε Νίλσεν, ε, ήμασταν ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Άντελφη, στην Επιτροπή Κοτέρ και τώρα ο κύριος Νίλσεν ρωτάει τι θα κάνουμε ε, για τα κράτη-μέλη και για να βελτιώσουμε τη συμμετοχή των περιφερειών. Και ρωτώ, σας το ανταποδίδω, εσείς τι κάνατε στη Σουηδία για να βελτιώσετε την κατάσταση, τι μπορούμε να μάθουμε εμείς από εσάς. Ε, βεβαίως και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική δομή. Σε όλα ε, τα κράτη-μέλη υπάρχουν ε, διαφορετικές διαδικασίες ε, λήψης αποφάσεων. Εκείνο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως θεσμός, όχι ως μεμονωμένα κράτη, είναι να βάζουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη, ε, το θέμα της ε, δέουσας ε, συμμετοχής του κατώτατου επίπεδου, το θέμα της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας. Και εμείς ως Επιτροπή των Περιφερειών το πράττουμε αυτό. Παραδείγματος χάρη, ξεκινώ με τα μεγάλα και τα διευρυμένα. Το θέμα, της τη συζήτηση για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση το διαδώσαμε και έτσι λοιπόν το θέμα αυτό συμπεριλαμβάνεται στο θεματολόγιο και μάλιστα έχει γίνει και αντικείμενο της επιστήμης. Επίσης, σε σχέση με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 εκφράσαμε το αίτημα να συνάπτονται οι περίφημες ε, εδαφικές συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη, όπου υπάρχει εγγύηση, προβλέπεται εγγύηση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που στήριξε αυτό το αίτημά μα Σε ορισμένα κράτη-μέλη μάλιστα σημειώθηκε πρόοδος επ' αυτού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επουδενή δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτά και μέχρι εκεί φτάνουν αυτά. Όσον αφορά τώρα στα διαρθρωτικά ταμεία και εκεί διαπιστώνουμε το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή την ε, συμπερίληψη ε, της τοπικής αυτοδικής και πάλι ανάλογα με το σύνταγμα που υπάρχει σε κάθε κράτος. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πιέζουμε για να μπει το θέμα στη μέση διάταξη. Στην Γερμανία λέμε έτσι χαρακτηριστικά ότι η πολιτική, όταν ασχολείται κανείς με την πολιτική, είναι σαν να προσπαθεί να τρυπήσει με το τρυπάνι έναν χοντρό και βαρύ τείχο. Η πολιτική είναι βαριά, είναι συμπιεσμένη. Εμείς όμως προσπαθούμε και νομίζω ότι σημειώνουμε κάποια μικρά βήματα. Θα ήθελα να από τον κύριο Μπόσνιακ να κάνει ένα σχόλιο και μετά θα περάσουμε ε, στο, στις επόμενες ερωτήσεις. Κοιτάξτε, εμείς αναμφισβήτητα στηρίζουμε τον κώδικα συμπεριφοράς. Αναμφίβολα υπάρχουν ε, αμφιβολίες και δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσον θέλουμε όλο αυτό το θέμα της εταιρικής σχέσης να το ξεκινήσουμε από το μηδέν. Γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Υπάρχουν αυτές οι επιτροπές ελέγχου οι οποίες σε περιφερειακό επίπεδο ασκούν κάποιες ε, αρμοδιότητες και αυτά στο πλαίσιο της εταιρική σχέσης. Άρα δηλαδή νομίζω ότι μπορούμε να προτείνουμε ένα μοντέλο ε, συμπεριφοράς προς μίμηση, αλλά η καλή αυτή εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει θα πρέπει να ε, τύχει περαιτέρω εκμετάλλευση. Επίσης, θέλω να σας πω, συμφωνώ ότι πρέπει να βρούμε μία συμβιβαστική πρόταση. Αφενός υπάρχει ο κώδικας, όπου ε, έχει τοποθετηθεί αρνητικά το Συμβούλιο, εγώ νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να αναζητήσουμε το συμβιβασμό και με αυτόν τον τρόπο να λύσουμε το θέμα. Ο κύριος Γκαρνιέ έθιξε ένα θέμα που αφορά στην υποστήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων. Το θέμα αυτό το εξετάσαμε οι μεγάλες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Δηλαδή, εκεί προβλέπεται οι μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν και αυτές τη δυνατότητα να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο. Αυτό βέβαια αφορά επιχειρήσεις οι οποίοι συνεργάζονται με μικρομεσαίες καταφεύγουν ε, στις δικές τους υπηρεσίες των μικρομεσαίων. Στόχος είναι να υπάρξουν αυτά τα κλάστερ τα επιχειρηματικά και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει πράγματι να υπάρχει η δυνατότητα και μεγάλες επιχειρήσεις να ε, λαμβάνουν υποστήριξη. Τώρα, όσον αφορά την κοινωνική οικονομία, και την ε, κοινωνική κατοικία. Αυτός είναι ένας ε, ιδιαίτερος τομέας. Η κοινωνική κατοικία πράγματι ε, πρέπει να την χάνει περαιτέρω υποστήριξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης πρέπει να βρούνε κάποια κονδύλια για την κοινωνική κατοικία, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να δημιουργηθεί εδώ ένα κενό. Για να λειτουργήσει βέβαια το όλο σύστημα ε, θα πρέπει να υπάρχει και ο απαραίτητος αριθμός ε, συνεργατών. Ε, κοιτάξτε, το θέμα της κοινωνικής κατοικίας είναι τελείως διαφορετικό στην Ολλανδία από ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη. Γιατί στην Ολλανδία το πρόβλημα είναι οι εταιρείε που κατασκευάζουν και τις κοινωνικές κατοικίες αλλά και τις ιδιωτικές κατοικίες. Άρα δηλαδή ε, εδώ τίθεται πραγματικά πρόβλημα δημόσιων ε, συμβάσεων και κρατικών ισχύσεων. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου η ε, Κομισιόν λέει ότι εκείνο που είναι καθοριστικό για τις κοινωνικές κατοικίες είναι το ύψος του μισθού. Αυτό όμως σας λέω αφορά τις κοινωνικές και όχι τις κρατικές κατοικίες. Συγγνώμη για την διακοπή. Τώρα, όσον αφορά τη στόχευση ε, από πλευράς ε, διαρθρωτικών ταμείων, στόχευση συγκεκριμένα θέματα. Έχουμε καλέσει ε, μέλη του Κοινοβουλίου να τοποθετηθούν πάνω στο θέμα, στο θέμα αυτό. Eh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βοσνιακά. Είμαι υπεύθυνο για τι εξωτερικέ ε, σχέσει ε, και για την ε, Γαλλική. Είμαι μέλο Επιτροπή κότερ τη Επιτροπή των Περιφερειών. Όπω καταλαβαίνετε, συμφωνούμε απόλυτα με την θεματική συγκέντρωση, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για την ανάπτυξη αντιγικής για την Ευρώπη του 2020 είναι αυτό. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να διερωτηθούμε και κάτι ακόμα. Ποια είναι η σχέση μεταξύ θεματική συγκέντρωση αφενός και μέλους, μέλου, μέλλοντό, συγγνώμη, τη αρχιτεκτονικής τη συνοχή στο τέλο, διότι δεν θα είναι το ίδιο το επίπεδο τη θεματική συγκέντρωση σε όλα τα θέματα, ανάλογα με του στόχου ε, και ανάλογα και ε, με, την, ε, με το σενάριο που θα ισχύει για την κάθε περιοχή στο 14 του 2020. Είναι ανοιχτό το διαπραγματευτικό κουτί. Στηρίζω το δίκτυο ασφαλείας, safety net στα αγγλικά, για περιφέρειες που βγαίνουν από το στόχο της σύγκλησης. Και δεν μιλάμε βέβαια για τον ενδιάμεσο μόνο στόχο, για τις περιφέρειες εκείνες που έχουν υπερβεί το ΑΕΠ δηλαδή έχει υπερβεί το 65% και φτάνει μέχρι το 9%. Μιλάμε για περιφέρειες που περνάνε το 85% του μεσόρου για πρώτη φορά. Ανεξαρτήτως ε, του ΑΕΠ που έχουν με αυτό με το οποίο βγαίνουν δηλαδή. Η Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη έκανε μια πρόταση, τη συζητήσαμε στην Επιτροπή μα και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ένα σαφέ μήνυμα στι κυβερνήσει για το διαπραγματευτικό κουτί. Ότι θα πρέπει να είναι δίκαιο και δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι τελικά εκπλήρωσαν ε, τι υποχρεώσει του. Και προχωρούν στην πραγματική σύγκληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ουλφ Βίκστρομ. Ορίστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι από το πρόγραμμα Interact που εδρεύει στη Φιλανδία του Τουρκού. Και εμεί ασχολούμαστε με την εφαρμογή της στρατηγικής για τη Βαλτική και θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να διασφαλίσει η θεματική συγκέντρωση τη στήριξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών γιατί αν έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες στα διάφορα προγράμματα μπορεί τελικά να καταλήξουμε να μην έχουμε κοινή στρατηγική ή προοπτική. με ε, εγώ θα ήθελα μονάχα να παρατηρήσω ότι ως εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, και να θυμίσω ότι όσον αφορά την ε, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση υπήρξαν ενστάσεις ότι στην πρόταση του κανονισμού δεν υπήρξε η αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στις κεντρικές κρατικές διοικήσεις από τη μια μεριά και τις αυτοδιοικητικές αρχές από την άλλη. Μάλιστα, ε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι κοινωνικοί εταίροι και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί αναφέρονται με μεγαλύτερη έμφαση, ενώ σε ορισμένε περιπτώσει μειώνεται ενοχλητικά ο ρόλο τη τοπική αυτοδιοίκηση και πολλές φορές αφομοιώνονται οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές στις, στην έννοια των κοινωνικών εταίρων. Ε, αυτά όσον αφορά την ε, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Τώρα για την ε, θεματική συγκέντρωση είναι θετική, κρίθηκε θετική από την Επιτροπή των Περιφερειών. Απλώς χρειάζεται να αμβληθεί ο σκληρός και ο περιοριστικός τρόπος με τον οποίο επιδιώκεται να επιτευχθεί. Dziękuję bardzo. Czekam na dalsze pytania w tym bloku. Czy ktoś z Państwa chce... Άλλοι παρακαλώ, επιθυμεί κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Dragi colegi, știm că agenda europeană privind simplificarea cadrului financiar... Αγαπητοί συνάδελφοι, η απλοποίηση του πολιετούς πλαισίου είναι κύριος πολιτικός στόχος και πρόκληση για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της απορρόφησης των κονδυλίων και να μειωθεί το γραφειοκρατικό άχθος. Η Κομισιόν έχει αρχίσει μία άσκηση επιτήρησης και βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα. Ξέρουμε λοιπόν ότι στόχος είναι να συνεχιστεί αυτό και μετά την εφαρμογή του κανονισμού θα ζητηθεί από τα κράτη-μέλη δηλαδή να κάνουν προσπάθειες απλοποίησης. Αυτό μάλιστα θα είναι ένα από τα κεφάλαια της, ε, των εταιρικών συμβολέων. Πώς βλέπει η Επιτροπή Περιφερειών, η Περιφερειακή Επιτροπή λοιπόν και γενικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ρόλο των τοπικών αρχών σε αυτήν την άσκηση απλοποίησης, το ρωτάω, γιατί σε όλες τις χώρες και στη Ρουμανία ανησυχούν πολλοί οι τοπικοί θύνοντες. Εμείς τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειών θεωρούμε ότι εφαρμόζοντας αυτά που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Δεοντολογία μπορεί να υπάρξει τεράστια απλοποίηση με πολύ θετικά αποτελέσματα. Πρέπει όμως να είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε τον κώδικα αυτών με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Κανείς άλλος. Θέλει κανείς άλλος το λόγο, όχι. Ε, τότε ίσως η κυρία Χιούμπνερ για τη στρατηγική της Βαλτικής. Ο, κοιτάξτε, ίσως θεωρήσετε ότι σας δυσκολεύουμε τη ζωή γιατί βάζουμε περισσότερες προτεραιότητες, περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης σε αυτό το πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας, αλλά απ' την άλλη μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Για την ερώτησή σας πώς θα διασφαλιστούν οι διαφορετικές αυτές προτεραιότητες ότι θα συνδυαστούν τελικά και θα υπάρξει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, αυτό στηρίζεται στο ότι από τις πρώτες φάσεις οι περιφέρειες που θα ήθελαν να συνεχίσουν τη συνεργασία της μακροπεριφερειακής στρατηγικής θα προσπαθήσουν ήδη από τότε να εφαρμόσουν μεγαλύτερη συνεργασία γιατί δεν είναι όλα τα προγράμματα τα ίδια ως προς τις προτεραιότητες. Μπορεί άλλα να έχουν περισσότερες δυνατότητες και να είναι συμπληρωματικά με άλλα. Αυτό που πρέπει να γίνει λοιπόν είναι να δούμε ότι η μακροπεριφερειακή στρατηγική πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συνεργασία και στη φάση των, συμβολέων, των εταιρικών συμβολέων και στη φάση της λειτουργίας των προγραμμάτων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος νομίζω για να διασφαλίσουμε τη συνεργασία γιατί δεν έχουμε χωριστό κεφάλαιο Επίσης πιστεύω ότι όλα τα μαθήματα που πήραμε μέχρι τώρα από τη στρατηγική της Βαλτικής δείχνουν ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί δεσμοί μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών που ήδη συνεργάζονται περισσότερο. Υπάρχουν περισσότερες συναντήσεις και το ανθρώπινο κεφάλαιο συνεργασίας ήδη υπάρχει. Άρα τα όλα αυτά τα προγράμματα μαζί μπορούν σε οποιοδήποτε τομέα τελικά να συνδυαστούν. Είναι παράδειγμα αυτό του πόσο αυτή η άτυπη, η soft συνεργασία και διαδικασία μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Επίσης όμως μπορούμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να κάνει σαφείς διαπραγματεύσεις με τις χώρες μέλη ότι για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές θα διασφαλιστεί τέτοιου είδους εμπειρία, γνώση. Θέλω επίσης να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή που έχω, που έχω το λόγο δηλαδή για να μιλήσω και για το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Δυστυχώς έφυγε ο ενδιαφερόμενος, αλλά το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται το βήμα-βήμα ή βήμα-βήμα διαδικασία δηλαδή απαιτεί μήνες για την προσαρμογή, αλλά πολλές χώρες μέλη ήδη έχουν ετοιμάσει τα συστήματά τους, τα εθνικά τους συστήματα προτεραιοτήτων και ήδη έχουν αρχίσει τις επαφές για τη συνεργασία που μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικές συμφωνίες συνεργασίας και εταιρικέ συμφωνίες και η Κομισιόν ήδη έχει αρχίσει να δημοσιεύει έγγραφα, πώς τα λένε, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα έγγραφα λέει η Πρόεδρος, αυτά τα έγγραφα για την κάθε χώρα. Άρα η συνεργασία μεταξύ χωρών και κομισιών έχει ήδη αρχίσει παρά το ότι δεν έχουμε ακόμη τον επίσημο κανονισμό. Είναι σημαντικό και αυτό γιατί αν περιμένουμε μέχρι να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις και να προετοιμαστούν τα προγράμματα τότε θα έχουμε πενταετή καθυστέρηση και γι' αυτό πρέπει να ξέρετε ότι να θεωρήσετε ότι τα όργανα θα κάνουν τη δουλειά τους, θα αποφασιστούν οι προϋπολογισμοί, εσείς απλώς να εγκρίνετε τα προγράμματά σας. Και τώρα για την απλοποίηση, τι μπορούν να κάνουν δηλαδή οι τοπικές αρχές για την απλοποίηση. Πάρα πολλά προβλήματα εθνικά και τοπικά δημιουργούνται. Μπορούμε και εμείς να βελτιώσουμε και στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν. Αλλά εσείς πρέπει να διαπιστώσετε να φροντίσετε να μην δημιουργούνται πρόσθετοι φραγμοί στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης πιστεύω ότι το πρωί ακούσαμε τον Έλληνα Υπουργό Ανάπτυξης που είπε ότι και αυτοί αρχίζουν την απλοποίηση. Βλέπετε ότι εθνικά υπάρχουν δυνατότητες απλοποίησης και αυτό πρέπει να γίνεται σαΐ αυτό είναι το καθήκον σας εσάς. Τώρα λοιπόν ε, θα ήθελα να ε, δώσετε το λόγο πίσω σε εσά. Θα περάσουμε πάλι στην εδαφική πολιτική. Την εδαφική διάσταση έχουμε το αστικό ζήτημα, ε, το urban, το έθισε ο Γιάν, την εδαφική διάσταση λοιπόν, αρχίζουμε να τη και βέβαια όλα αυτά αφορούν τη συνεργασία, τοπική ανάπτυξη, την αστική ανάπτυξη, αλλά και τα νέα εργαλεία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε το τοπικό επίπεδο, πώς να το πω, να κινητοποιηθεί, να δραστηριοποιηθεί και να συμμετάσχει ενεργά στην πολιτική. Αγροτική ηθικό, ε, Άστη, είναι ζητήματα διάφορα αυτά. Η μεταφική διάσταση πρέπει να ενισχυθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια, ανησυχίε, ή ερωτήσεις. Κύριε Όσφαλ, θέλετε το λόγο. Ναι, όχι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ο εισηγητής για την εδαφική συνεργασία και για την εδαφική συνοχή. Νομίζω λοιπόν αυτή η εδαφική διάσταση είναι πραγματικά σημαντικότερη για την συνεργασία. Το θέμα δεν είναι να εφαρμόσουμε τη στρατηγική 2020 ε, θα πρέπει να υπάρχουν και προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της ε, στρατηγικής. Διότι αν περιοριστούμε μόνο σε ορισμένα θέματα, τότε ε, θα έχουμε κατά κύριο λόγο μόνο την κουβέντα για την έρευνα και την ανάπτυξη. Και δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να συζητήσουμε για διάφορες προϋποθέσεις και να τις συνδέσουμε μεταξύ τους. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει. Όταν μιλάμε για τον τουρισμό, να στηρίξουμε τον τουρισμό. Ε, όσον αφορά τη στρατηγική για τη Βαλτική, η στρατηγική αυτή προέκυψε ακριβώς στη Βαλτική και περιλαμβάνονται ε, εκεί οι εκτάσεις ε, που αφορούν την περιοχή δεν επιβάλλεται τίποτα από τα πάνω. Αυτές όμως ε, οι περιοχές είναι πολύ διαφορετικές και αν δούμε λιγάκι τη στρατηγική για τον Δούναβη υπάρχουν μεγάλες πόλεις, υπάρχουν τουριστικές και φτωχές ε, περιοχές κάθε περιοχή χρήζει διαφορετικής ε, προσέγγιση. Ο στόχος της μακροστρατηγικής έγκυται στο ότι προέκυψε μάλλον διότι ε, αυτοί που τον ε, εκπώνησαν θέλησαν να έχουν ένα σύνολο ε, με διαφορετική βέβαια προσέγγιση. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να υπάρχει πολύ στενή αλληλένδεση. Ο Γιάννη Όλμπριχτ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες σύντομα, αν με επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα έχουμε κάποια στοιχεία στον κανονισμό και κάποια στοιχεία στην πολιτική προσέγγιση. Για παράδειγμα, στην πολιτική προσέγγιση, τι έχουμε. Μακροπεριφερειακή στρατηγική. Εδαφικό είναι αυτό. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν υπάρχουν κονδύλια για αυτή τη διάσταση. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Περνάνε από τα project, από τα έργα τα χρήματα. Δεύτερον, το πρόβλημα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Τελείως δύο διαφορετικές πολιτικές. Ναι, ναι, ναι στα χέρια δύο διαφορετικών εντελώ μεταξύ του Υπουργείων. Για πρώτη φορά, για πρώτη φορά επαναλαμβάνω, έχουμε κοινό προγραμματισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν το έχουμε στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο, το CSF, τα είπε και ο Μάρικ Βόζενκ πριν, θα το έχουμε και στην εταιρική σχέση και τη σχετική σύμβαση. Άρα απαιτείται συνεργασία μεταξύ ανθρώπων από την πολιτική γεωργία και ανθρώπων από την πολιτική συνοχή. Θέλω λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σα στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει τώρα το εγχειρίδιον για τη συνεργασία μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών. Τον επόμενο μήνα στο ΜΕΣ θα γίνει η πρώτη συνάντηση, στη Βαρσοβία την άνοιξη δεύτερη και ίσως η τρίτη στις Βρυξέλλες. Και θα είναι έτοιμο λοιπόν έτσι το εγχειρίδιο για τη συνεργασία μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Σας το λέω για να το ξέρετε, γιατί ναι. αυτές είναι εξελίξεις. Τρίτο στοιχείο. Το περίφημο 5% του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του ΕΤΠΑ. Υπήρχαν κάποιες φήμες ε, ότι το 5% πάει στις πόλεις. Λάθος. Το εξεργαζόταν και η Επιτροπή των Περιφερειών. Όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε, δεν μιλάμε για 5% πάει στι αλλά ένα πιλωτικό σχέδιο για τα κράτη-μέλη που πρέπει να προετοιμάσουν το πρόγραμμα για τις πόλεις και τα περιχωράει του γείτονες. Όχι όμως 5%. Και ούτε υπάρχει όριο στα επιχειρησιακά προγράμματα για τις πόλεις. Το 5% αφορά ναι. αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Αυτά είναι τα εδαφικά στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά. Και αν με επιτρέπετε άλλη μια παρατήρηση. Γιατί είπε ο συμπρόεδρος ότι είναι συναφή τα έγγραφα του Επιτροπή των Περιφέρων και του Κοινοβουλίου. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Oh. Γιατί έχουμε του ίδιου στόχου. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και επειδή συνεργαζόμαστε είναι παρόμοιε οι θέσεις μας. Ευχαριστώ.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 να σας πω κάτι σχετικό με αυτή τη στρατηγική. Έχω συζητήσει το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ροή ενημέρωσης για τη στρατηγική αυτή και πώς μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά οι εταίροι μας στρατηγική αυτή. Χρειαζόμαστε καλύτερη ενημέρωση και διάφορες δράσεις για να βελτιώσουμε τη στρατηγική αυτή. Η ροή πληροφοριών και ενημέρωσης μεταξύ κρατών και εντός κρατών πρέπει να βελτιωθεί. Γιατί έτσι θα μπορούν όλοι να δεσμευτούν περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία. Καλ Σνάιντερ. Καλή Σνάιντερ. Ja, danke. Ich würde gerne... Äh, Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ έτσι λιγάκι γενικότερα σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Ολμπρίχτ. Έχω την αίσθηση ότι η συζήτηση σήμερα δεν ε, είναι αρκετά ζωντανή διότι το θέμα το έχουμε συζητήσει πολύ κατά το παρελθόν, ε, καταλήξαμε σε κοινέ θέσει. και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους όλων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ότι μπορούσαμε, μας δόθηκε η δυνατότητα στο παρελθόν να έχουμε αυτή την έντονη συζήτηση και τότε προέκυψαν πάρα πολλές απόψεις που ακούστηκαν. Αν θέλετε τώρα είμαστε σε στάση αναμονής. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο Συμβούλιο, τι θα γίνει το Νοέμβρη, ποιες αποφάσεις θα ληφθούν για το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και ποιες ε, θα είναι επιπτώσεις στους διάφορους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία. Τις, ε, τα τελευταία δύο χρόνια έχω πει επαν, επανειλημμένα ότι εγώ χαίρομαι και χαιρετίζω το γεγονός ότι η συνθήκη της Λισαβόνας <coughs> εκχωρεί περισσότερα ε, δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα μάλιστα συνειδητοποιώ πόσο τυχεροί είμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει αυτά τα επιπρόσθετα δικαιώματα. Γιατί προφανώς ε, κανείς μας δεν θεωρεί ότι ε, στο Συμβούλιο θα είμαστε ικανοποιημένοι με τις αποφάσεις ε, για το δημοσιονομικό πλαίσιο και οτιδήποτε άλλο. Πόσο καλό λοιπόν είναι που συναποφασίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι εταίρος μας στις διαπραγματεύσεις. Το λέω αυτό ξεκάθαρα. Εμείς θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ε, ο δικηγόρος με τη δική μας την πλευρά, με τα συμφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης και γι' αυτό θέλω να πω ότι η συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα πραγματικά άξιζε τον κόπο. Βεβαίω, ελπίζω ότι αν τελικά χρειαστεί να υπάρξουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις θα παίξει βέβαια η πολιτική συνοχή σε κάποιο ρόλο, όπως, όμως και πολλά άλλα θέματα. Σε αυτές λοιπόν τις διαπραγματεύσεις να καταστεί σαφές τι ακριβώς σημαίνει όταν οι ε, διαπραγματεύσεις καρκινοβατούν. Γιατί όταν καρκινοβατούν αυτό σημαίνει για μας στις ε, περιφέρειες ότι δεν θα μπορέσουμε την 1η του 14 να έχουμε καταρτήσει τα λειτουργικά μας προγράμματα, άρα δηλαδή δεν θα μπορούμε να επενδύσουμε κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων θα προκύψει ένα κενό και αυτό το κενό σίγουρα δεν θα βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση. Γι' αυτό λοιπόν Παρακαλώ να μην φυστείτε ούτε κόπου ούτε χρόνου σε σχέση με τις ε, νέες διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν. Πολύ ωραία. Κλείνουμε λοιπόν αυτά τα θέματα. Μισό λεπτό. άλλο ένας έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much. Uh, from Ευχαριστώ από το EuroCities θα θέλαμε το Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξουν την ε, ανάθεση ε, της χρηματοδότησης ε, στις πόλεις. Πολλοί θα ήθελαν, πολλές πόλεις θα ήθελαν να υπάρξει αυτή η εκχώρηση αρμοδιότητας, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε σε τοπικό επίπεδο, να δώσουμε μεγαλύτερη ορατότητα, ιδιοκτησία αν θέλετε, και να υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση σε τοπικό επίπεδο. Είναι προαιρετικό ή μήπως απλά θα ήταν τελικά και συμμετοχή στην επιλογή των, πόλε, των ε, project, δηλαδή να συμμετέχουν οι πόλεις. Αυτό δεν θα μας ε, φαινόταν και σωστό. Θα ήθελα να σας απαντήσω. Η απάντηση δεν είναι μόνο στα χέρια του Κοινοβουλίου, η απάντηση είναι και στα χέρια των περιφερειών. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα της εκχώρησης ε, της ε, διαχείρισης, ακριβώς αυτό που μόλις τώρα είπατε, αφορά στο περίφημο ε, τουλάχιστον 5%. Αυτό δεν είναι πρόβλημα προγραμμάτων, είναι πρόβλημα όχι projects, αλλά πρόβλημα προγραμμάτων. Το Κοινοβούλιο για 7 χρόνια αποφάσισε να εκχωρήσει αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά οι κυβερνήσεις και οι περιφέρειες αντέδρασαν. Δεν θα τις κατονομάσω αυτές τις ε, περιφέρειες, αλλά εν πάση περιπτώσει είπαν ότι οι πόλεις δεν είναι έτοιμες να κάνουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση του Κοινοβουλίου προσφέρει τη δυνατότητα να λαμβάνεται προαιρετικά η απόφαση. Είτε όλη η αντιπροσωπεία είτε κάποιοι, μερικοί που επιλέγουν τα προγράμματα, τα ελέγχουν και το καθεξής. Δηλαδή, η δική μας η αντίδραση είναι να προτιμήσουμε το ευέλικτο σύστημα το οποίο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν να αποφασίσουν τι, να αποφασίσουν αν θα εκχωρηθεί η διαχείριση των προγραμμάτων στις πόλεις ή όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε αισιόδοξοι. Την τελευταία φορά, πριν από 7 χρόνια, προτείναμε τη διαχείριση να την αναλάβουν οι πόλεις και ε, πολλοί αρνήθηκαν κατηγορηματικά, απορρίφθηκε μάλλον αυτό, λόγω της επικουρικότητας. Δεν σημαίνει όμως τώρα το ίδιο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πάντως, ε, και τελευταία μου παρατήρηση, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις πόλεις απαιτεί πολύ στην συνεργασία με τις περιφέρειες. Αν οι περιφέρειες διαπιστώσουν ότι οι πόλεις είναι έτοιμες, τότε το όλο πρόγραμμα θα προχωρήσει. Αλλά ε, εντωμεταξύ είναι απαραίτητο να υπάρξουν δύσκολες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις περιφέρειες και τις πόλεις. Πάντως πιστεύω ότι ακόμα και μία μερική εκχώρηση θα αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός. Πολύ ωραία. Εγώ ω εκπρόσωπος ε, περιφέρειας ε, θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω η συνεργασία ανάμεσα στις πόλεις και τις περιφέρειες σε πολλές περιπτώσεις ήταν πολύ καλή και πολύ υποφελής για τις ε, πόλεις. Τώρα, όσον αφορά τα κονδύλια, η όλη συζήτηση είναι ακόμα ανοιχτή. Ας πάμε τώρα ε, στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Η συγητής ε, ως εισηγητής ε, της ε, Επιτροπής, αρμόδια Επιτροπής, θέλω να πω το εξής. Της Επιτροπής των Περιφερειών, θέλω να πω το εξής. Έχουμε μια κατεξουσιοδότηση πράξη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή την πήραμε ω βάση. Τώρα όμως η κατάσταση έχει αλλάξει. Η Επιτροπή έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά μας και συνεργαστήκαμε στενά με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών. Η κατάσταση λοιπόν είναι η εξής. Αφενός ε, έχουμε κάποιες ρυθμίσεις στο παράρτημα. Ε, κατά τα άλλα, όσον αφορά της, ε, την πραγματική νομική πράξη, έτσι συμφωνήθηκε τουλάχιστον, έχουμε την κυρία Φανκρέλ και τον κύριο Φανίστελ Ρόι, οι οποίοι συνεργάστηκαν στενά. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή ε, θα προτείνει ε, εξουσιοδότηση πράξη που θα αφορά στις εταιρικές ε, συμβάσεις. Θα υπάρχει έτσι μια παράλληλη εξέλιξη. Θα έχουμε το παράρτημα και θα έχουμε και ένα επιπρόσθετο έγγραφο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι όλα αυτά αποτελούν βελτίωση γιατί πλέον έχουν αρθεί ε, κάποιες λήψεις. Ε, τώρα στο άγγραφο γίνεται λόγος για ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή διατύπωση και πέραν αυτού υπάρχει και ένας κατάλογος, ενδεικτικός κατάλογος παραδειγμάτων προς μίμηση ε, και έτσι θα είναι δυνατόν να γίνει και κάποια επιλογή. Αυτή την κατεύθυνση ακολουθούν οι εργασίες στις ε, συζητήσεις ανάμεσα στη δική μας την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπάρξει ε, κάποια συμφωνία και εάν μου επιτρέπετε εμείς είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Βεβαίως και θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Παρόλα αυτά όμως πρόκειται για έναν καλό συμβιβασμό εφόσον μιλάμε για ένα κοινό ε, στρατηγικό πλαίσιο. Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρξει ταχεία έγκριση αυτών των νομικών πράξεων. Παρότι βέβαια ε, θα μπορούσε κανείς ε, ε, να θέλει να προχωρήσουν τα πράγματα γρηγορότερα. <clears throat> Για αυτή τη στιγμή υπάρχει χρονική υστέρηση. Μήπως έχετε κάτι να πείτε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά αν θέλετε κάτι να πείτε υπάρχει λίγος χρόνος. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιος το λόγο, κανείς δεν επιθυμεί το λόγο, άρα δηλαδή, ε, α, μισό λεπτό, ε, κάποιος ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να είμαστε πλήρεις. Δυστυχώς ο συνάδελφός μου πρέπει να φύγει για να πάρει το αεροπαλάνο, αλλά αφού είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, όχι απαραίτητος των πόλεων αλλά και το, της υπαίθρου και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ίσπραξη των κοντιλίων όχι μόνο των περιφερειακών βλέπουμε και εμείς ότι στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο πρέπει να διασφαλιστεί όποτε είναι δυνατόν να διατίθενται τα κονδύλια κατευθείαν στις τοπικές αρχές. Καμιά φορά βέβαια δεν γίνεται τεχνικός, αλλά σε άλλες περιπτώσεις γίνεται. Τονίζω απλώς την ανάγκη να μην κοιτάζουμε μόνο το θέμα των πόλεων, αλλά γενικά να μιλάμε για τοπικές αρχές και κοινότητες. Σε μερικές χώρες μέλη, που είναι πολύ χαμηλά τα ποσά που διαθέτει το κράτος, μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό το συμπλήρωμα από την Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που συζητήθηκαν αυτά τα θέματα. Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι αυτή η γνωμοδότηση θα ληφθεί υπόψη. Δεν έχουμε πια αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα σιγά σιγά να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση. Νομίζω ότι οι επαφές ε, ανάμεσα στην Επιτροπή των Περιφερειών και την Γενική Διεύθυνση, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Επιτροπής είναι πολύ καλές και νομίζω αυτή η συνεργασία έχει οδηγήσει ε, στο μέλλον ε, να συντάσσονται έγγραφα τα οποία θα προάγουν την περαιτέρω συνεργασία. Αυτά τα οποία είπατε σήμερα το πρωί θα προσπαθήσουμε να τα συμπεριλάβουμε στις δηλώσεις της Επιτροπής των Περιφερειών. Όλα αυτά θα έχουν προετοιμαστεί μέχρι το τέλος του έτους. Γι' αυτό λοιπόν ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, σκέψεις που εκφράσατε. Ε, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε <clears throat> αυτή τη συνεργασία και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ και δίνω και πάλι το λόγο στην Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Να κάνω ένα σχόλιο για το... την παρέμβαση από το EuroCities Θυμάμαι το 2005, το 2006, όταν ε, ήμουν στην Κομισιόν, τότε ήμουν επίτροπο και τότε δεν μπόρεσε να υπάρξει αυτή η δυνατότητα εκχώρηση των Δεν ξέρω τι έγινε στο μεταξύ και αν κάποιο κατάφερε να το κάνει. Πρέπει να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τώρα για να καταλήξουμε όμως, χαίρομαι πάρα πολύ μέσω Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, γιατί καταφέραμε να έχουμε αυτή τη συνεργασία τα τελευταία χρόνια με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Κότερ, της Επιτροπής των Περιφερειών, που έρχονται με προτάσεις, με γνωμοδοτήσεις, ε, έχουμε ανταλλαγή απόψεων, ε, μας ακούν, τους ακούμε και με αυτή την προσέγγιση μπορούμε να επηρεάσουμε πραγματικά Γιατί... δεν πειράζει, ε, ξέρω, 999 δολάρια, ναι, ναι, Είναι καλό να μπορούμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον. Συμφωνώ με όλους όσους λένε ότι ακόμη και το καλύτερο δυνατό νομικό πλαίσιο δεν μπορεί να κάνει τίποτε αν δεν υπάρχει ένας εξωπρεπής προϋπολογισμός. Αυτή είναι η πρόκληση για μας ιδίω. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ σημαντική πρόκληση και εσείς όμως θα πρέπει στις χώρες σας με τις κυβερνήσεις σας να δείτε τι μπορείτε να κάνετε γιατί οι πρωθυπουργοί σας, οι κυβερνήσεις σας έχουν αυτή την ιδέα να είναι ως το τον πιο μικρός ο προβλησμός. Εντάξει, όχι όλοι, αρκεί ένας να πει όχι και δεν χρειάζεται και δεύτερος. Λοιπόν, παρακαλώ κάνετε και εσείς λίγο λόμπι στις χώρες σας και θέλω να πω και κάτι ακόμη. Βλέπουμε αυτή την περίοδο που πραγματικά πρέπει ε, να περιοριστεί ο εθνικός προπολογισμό επί των κρατών μελών Τρει φορές κοιτάμε πού επενδύουμε το κάθε ευρώ. Απόλυτα θεμητό είναι λοιπόν και οι κυβερνήσει να βλέπουν πώ επενδύονται και τα χρήματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και κάποιε φορέ του διαφεύγει ότι υπάρχουν κάποιες αρμοδιότητες που μπορούν να συνδεθούν με αυτούς τους πόρους. Ίσως υπάρξει τάση να υπάρξει εκ νέου συγκέντρωση, ενώ εμείς είχαμε πετύχει αποκέντρωση σε κάποια επίπεδα. Πρέπει να είστε λοιπόν προσεκτικοί να επαγρυπνείτε για να μην χάσουμε τα κεκτημένα μας και να δούμε και τι μπορούμε ακόμη περισσότερο να πετύχουμε παίρνοντα στο πλευρό μας σε αυτή την προσπάθεια το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Πάρτε το σοβαρά λοιπόν και μην επιτρέψετε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ολοκληρώνω με αυτό. Έχω όμως και μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Όσοι δεν ανήκουν σε Επιτροπή Ρέτζι το κοινοβούλιο πρέπει να φύγουν τρέχοντας από την αίθουσα. Γιατί έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες και δυστυχώς πρέπει να βιαστούμε. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που σας παρακαλώ να φύγετε όσο το τον πιο γρήγορα από την αίθουσα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά πάντως. Okay, please. Okay, secure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 I would like to start the vote. Αρχίσουμε τις ψυχοφθορίες τώρα. Και οι συντονιστές και οι συντονίστριες τουλάχιστον να έρθουν εδώ στη μέση να τους βλέπω. Για να έχω μια ιδέα. προτιμάς εκεί στην άκρη, μα δεν μπορώ να σε βλέπω από εκεί, ε, παιδί μου. Σχεδόν έτοιμοι είμαστε και έτοιμες για να αρχίσουμε τις ψηφοφορίε. Βάλατε, φέρατε τις κάρτες σας. Αρχίζουμε την ψηφοφορία για την έκθεση Μανέσκου, τροπολογία 61. Δεν είπαμε υπέρ ακόμα, 61. Λοιπόν, τι ξανά, μας παρακαλώ. Για να αρχίσουμε λοιπόν. Τροπολογία 61 υπέρ Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 62 επομένως υπέρ. Κατά. Κατά. Απορρίπτεται. 63 και 64 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται 65 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω. Επαλήθευση για την 5. Επαλήθευση. The vote is open. The vote um, is closed. Yeah. Πάει, έληξε. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Ποιες. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απαρρίπτεται 67 υπέρ κατά Ποιες; απαρρίπτεται 68 υπέρ κατά Ποιες; Ρίπτεται. 69 υπέρ κατά Ποιες; ρίπτεται 70 υπέρ κατά Ποιες; εγκρίνεται 8 υπέρ κατά Ποιες; εγκρίνεται 73 και 74 υπέρ. Κατά. Yes. Απορρίπτονται. 75 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 76 και 77 υπέρ. 76 και 77 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 78 και 79 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 9 υπέρ. Α, έχει καταπέσει. Α, μάλλον 9, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 και 87 υπέρ κατά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 17 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 18 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 19 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 20 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 93 υπέρ, κατά, χες, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, όχες, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, όχες, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά ποιες εγκρίνεται 27 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 28 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται όχι 28 Απαλήθευση για την 28 γιατί έχει αμφιβολίες ο Μιγγέλ εγκρίνεται καλά τα είπα συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ, συμβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 98 δεν ψηφίζουμε 102 υπέρ, κα, υπέρ, υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται 103 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108, 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113. 113 δεν έχει αποσυρθεί υπέρ. 113 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. «32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 115 και 16 υπέρ, όχι, α όχι, γιατί εγκρίθηκε η 32 λοιπόν. 117 και 118 υπέρ, κατά ποχές απορρίπτονται, 33 υπέρ, κατά ποχές εγκρίνεται, 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 119 και 120 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται, 120 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 122 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 και 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 131 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 132 υπέρ κατά αποχές είπα 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 45 υπέρ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 αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά έληξε 32 υπέρ 7 κατά μία αποχή εγκρίνεται τώρα η έκθεση του Όλτριχ Βλάσακ για τον αριστικό προστασία 50 υπέρ. Κατά. Τι, πώ, πώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ. Ω επαλήθευση για την 50, γρήγορα όμω γρήγορα, γρήγορα. Έληξε. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για την 51. Επαλήθευση. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Για την 53 χρειάζεται απαλήθευση. Ξανά για την 53 ηλεκτρονικά. 53. Έληξε. Απορρίπτεται πανηγυρικά. Και δεν το είδα. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Θέλετε παλήθευση την 55. Ω Θεέ μου. Παληθεύεται. Έλξε. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο. 55 υπέρ. Άμα δεν μου τα λέει ο συντονιστής πρέπει να ξαναμετράω κάθε φορά λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ της 55 ξανά. Εγκρίνεται, ορίστε. 56 υπέρ. Κατά. Αγιές, απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αγιές, εγκρίνεται 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 63 υπέρ είπα 63 υπέρ οι φιλελεύθεροι δεν ψηφίζουν 63 είπαμε 63. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 64. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος επαλήθευση για την 65. Απορρίπτεται με ισοψηφία. 66 υπέρ Κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. ...67 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται 71 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, επαλήθευση για την 72 έληξε εγκρίνεται με μία ψήφο 20-19 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ, κατά αποχές Νομίζω απορρίπτεται. Επαλήθευση για την 80. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 81 και 82 υπέρ. Κατά. Οχές εγκρίνονται. ψηφίσαμε αδίκως. 83 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 84 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 85 υπέρ, επαλήθευση για την 85. Έληξε. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται Επαλήθευση. Α, το ήξερα. Επαλήθευση. Άμα δεν εγκρίνεται ο Μάρκος μου ζητάνε πάντα επαλήθευση. Απορρίπτεται Μάρκο μου. 92. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Νομίζω πάλι είναι ασαφές. 92 επαληθεύεται. Έληξε, απορρίπτεται με μία ψήφο. 93 υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται 94 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται 20 Α, έχει αποσυρθεί 96. 96 υπέρ. 96. Αποχές, αλλά δεν Α, επανήθευση, επανήθευση. Ε, ξέρω, ξέρω, θέλετε επανήθευση. Για να ξέρετε πώς θα ψηφίζουμε, τέλος πάντων. 96 επαληθεύεται. Α, ξέχασα να ψηφίσω και η ίδια. Απορρίφθηκε. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά νομίζω απορρίπτεται μπορούμε αν θέλετε να ελέγξουμε την 99 την ελέγχουμε εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ Α, επαλήθευση για την 103 104 εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επαλήθευση την 22. Έληξε, απορρίπτεται με ισοψηφία. 105 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται νομίζω. Μάρκο θέλεις επαλήθευση, 105 επαλήθευση. εγκρίνεται με μία ψήφο. 106 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές. Αν θέλεις να ελέγξουμε Μάρκο, εγώ βλέπω ότι απορρίφθηκε, αλλά μετά θα μου πεις έλεγχο, έλεγχο. Εγκρίνεται με μία ψήφο. στενά τα όρια. 108 υπέρ. Έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί μεταξύ ομάδων γιατί πολλοί απουσιάζουν. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε από τις ομάδες απριόρι. 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. τώρα 116 μου λένε. 116 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. σε επαλήθευση μάλιστα. 116. Απορρίφθηκε. 117 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται Μάρκο και από τους δικούς σου. Δεν ελέγχω λοιπόν. 118 κατά αποχές. Απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται και τώρα 24 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 1 υπέρ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 Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. 34 υπέρ. Α, έχει καταπέσει μάλιστα, μάλιστα. 35 υπέρ, κατά, ποχές, απορρίπτεται. Έλα παιδί μου, δύο ομάδες υπέρ και μία αποχή, 36 υπέρ, κατά, αποχές, αγκρίνεται, 37 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά δεν χρειαζόταν να ψηφίσουμε μάλιστα μάλιστα μάλιστα 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ επαλήθευση της 7. Ισοψηφία απορρίπτεται. Πού να το ξέραμε. Απορρίπτεται ορίστε. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 8 έληξε απορρίπτεται 9 γιατί 48 έχει αποσυρθεί 9 υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται θέλεις επαλήθευση όχι όχι ρε παιδί μου ε, Ελέγξαμε τόσες φορές για τον Μάρκο που άση τώρα. Δεν ψήφισαν όλοι, τι να κάνουμε. Έληξε ψηφοφορία, εγκρίνεται. Τώρα το σύνολο του κανονισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Ο κύριος Αυγίας. Το αποτέλεσμα. 34 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. Τώρα, τώρα λέγω η έκθεση του κυρίου Αυγία. Είναι το σημείο 11 της μερίσιας διάταξης. Χρηματοδότηση, διαχείριση και υπάρκωση της κοινής πολιτικής. Άλλο έχω εγώ. Δεν ξέρω. Ωραία, λοιπόν, τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, γκρίνεται. Τροπολογία 7, αποχές, εγκρίνεται. 8. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 37 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, ε, κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Όχι, 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Τι κάνουμε, τι κάνουμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, 18 υπέρ 19 Κατά λοιπόν, πάμε 42, απορρίφθηκε η προηγούμενη. 42 εγκρίνεται, 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 48 μη παραδεκτή. 14 υπέρ. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος έλεγχος για το 14. Μπορεί και να έχετε και δίκιο. Απορρίπτεται, ναι. Μάλιστα. Απορρίπτεται το 14. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πού πάμε τώρα, στην 20. 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ρισάει τα αστεολογικές σκέψεις δηλαδή. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Όχι, έχει απορριφθεί, αποσυρθεί, συγγνώμη. Πού πάμε, στη συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Να ελέγξουμε κατευθείαν 33 λέω. Ελέγχουμε. Άρχεται, πέραση ψηφοφορίας, εγκρίνεται και τέλος 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα συνολικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ωραία. Μόνο δύο απέσχων. Περνάμε τώρα στην έκθεση της Κατρίν Γκρες. για τις άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθετών στήριξης της ΚΓΜ. Λοιπόν, 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Νομίζω, έλεγχος Ελέγχουμε την 11. Ελέγχω. Πέρασε. Εγκρίνεται. 22 προς 18. Πάμε τώρα. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά, αποχές, ελέγχουμε. Ελέγχουμε τη συμβαστική 1. Mm. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεκαπέντε. Α, απορρίφθηκε η συμβαστική ένα. Ναι, 50 τότε. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά απορρίπτεται. 15 τώρα υπέρ κατά απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Εντάξει, να ελέγξουμε. Μη και διστάσω, ορμάτα αμέσω. Ναι. Λοιπόν. 21 υπέρ, 19 κατά εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Το ίδιο νομίζω είναι, αλλά ας ελέγξουμε και τα 17. Απορρίπτεται. Μισοψηφία. 20 όλα. Τροπολογία 19. Προφορική τροπολογία είναι κάποιο κατά τη τροπολογία του κ. Σικέρη. Και στο χέρι του, άρα δεν ψηφίζουμε. Τι δεν ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε την προφορική. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία χωρίς την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Ελέγχουμε. Ε, 19. Χωρίς την προφορική. Δεν ψηφίζει κανένα. Τι γίνεται. Λοιπόν, εγκρίθηκε τελικά με μία ψήφο διαφορά. Να ξαναελέγξουμε. Τι πρόβλημα υπάρχει, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να μιλήσω εκ μέρους της εισηγήτριας της γνωμοδότησης μας, αυτής της κυρίας Κατρίν Γκρέζ, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ. Κυρία Γκρέζ, εκφράζει την λύπη της για την αντίθεση του ΕΛΚΑ στην προφορική της τροπολογία, που αποτέλεσε καρπό συμβασμό των ε, σκιώδη εισηγητή της Άλτων, κυρία κύριο για αυτό το θέμα που αφορούσε την πρόταση να υπάρχουν κάποια εδαφικά σύμφωνα ε, μεταξύ των κοινωνικοπικληματικών εταίρων και των τοπικών πολιτικών για την εφαρμογή πράσινων πρακτικών που θα λαμβάνουν υπόψη τα εδαφικά χαρακτηριστικά. Η πρόταση αυτή αρχικά προέρχεται από την Επιτροπή των Περιφερειών. Κυρία Κρέη, σας ενθαρρύνω να ψηφίσετε την αρχική, τις αρχικές τροπολογίες, δηλαδή 3 και 19 γιατί αυτό θα δώσει ένα σημαντικό μήνυμα ότι δηλαδή εμείς θέλουμε να ληφθούν περισσότερο υπόψη και να εισακουστούν καλύτερα οι εδαφικοί εταίροι. You Μήπως θέλετε να ξανα, ξαναψηφίσουμε, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι συμβιβασμός, αλλά ψηφίσαμε. Να μην επανέλθουμε. Ευχαριστώ που το ζητάτε πάντως, αλλά... Λοιπόν, τότε πάμε στη 18, λέει πρόεδρος. Εντάξει, ψήφι υπέρ της 18. Ναι. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 55, όχι, μην παραδεκτεί. 56 υπέρ. 56 υπέρ. Κατά αποχές, ναι, ναι, νομίζω απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 22. Is... Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Και πού πάμε. Στην 64. 64. Ε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 68 ναι, ναι. υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 27. απορρίπτεται 21 προς 18. Τροπολογία 30. Δεν την έχω εδώ. Α, την είδα. 30. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλω να ελέγξουμε, ελέγχουμε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32 υπέρ, κατά αποχές. Πάρα πολύ αμφίροπο. Πάλι δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Να ελέγξουμε το 32 παρακαλώ. Mm. Απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, νομίζω, 85 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τεολογικές σκέψεις, συμβιβαστική 2, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 36 όχι, ναι, 36 υπέρ, κατά, ποχέ. εγκρίνεται. Ναι. Ας το ελέγξουμε καλύτερα, 36. Έχω μπερδευτεί. Ελέγχουμε λοιπόν τέρμα, έλλειψη ψηφοφορία, εγκρίνεται. Ναι. Η 36. Καταπίπτει 35 επομένω. Πάμε στην 37. Ψήφι περ. Κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται. 39 υπέρ. 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 τώρα με προφορική τροπολογία. Είναι κάποιος αντίθετος στην προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποιο που είναι αντίθετο. Άρα ψηφίζουμε χωρί την προφορική τροπολογία την τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχέ, νομίζω εγκρίνεται. Ή να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε, ελέγχουμε. προς 19 εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω με την ίδια διαφορά ψήφων. Να ελέγξουμε, ελέγχουμε. Ναι. Ελέγχουμε 42. Ναι, ελέγχουμε. Ναι, Απορρίπτεται μισοψηφία. Πάμε τώρα στη 43. Υπέρ. Υπέρ. Εγκρίνεται νομίζω. Να ελέγξουμε θέλετε και τη 43. Ας την ελέγξουμε. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20 προς 17. Τελική ψηφοφορία, με το σύνολο τώρα, νομοδότηση. Ηλεκτρονικά. Why we It's adopted, right? Yes. How we calculate it? 18 to 4 against and... 18 υπέρ 4 κατά και 17 αποχές. Περνάμε τώρα στην επόμενη Γιουνούς Ομαρζή, ο συντάξης γνωμοδότησης. I'm supposed to say. Λοιπόν, συμφώνησε ο συνάδελφος ως εισηγητής να πάρει ε, κάποιες τροπολογίες πίσω και έτσι έχουμε διευκολύνει κάπως τα πράγματα, αλλά ξεκινάμε στη δεύτερη σελίδα με την 33 τροπολογία, πέρα κατά αποχές συγκρίνεται. Πηγαίνουμε μετά στην 37 που έχουμε μία Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές Τροπολογία 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, δεν ξέρω τι γίνεται. Μου κάνει τη ζωή δύσκολη η ECR. Για να ελέγξουμε παρακαλώ τη 40. 41, απορρίφθηκε 40. 41, ε, υπέρ, κατά. Το ίδιο πράγμα. Νομίζω απορρίπτεται. Να μπορούμε να το ελέγξουμε όμως για να επιβεβαιωθεί. 41, ελέγχουμε. Πράγματι απορρίπτεται. Πάμε. Πάμε. Πού πάμε. Στην 68 σελίδα 4 πάμε. Υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. με μία ψήφο περίφθη. 69 υπέρ, κατά αποχές, Πάμε τώρα σε τολικέ σκέψει του στο recital. Στην τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα σε 15 υπέρ, κατά. Α, εγκρίνεται νομίζω. Όχι, δεν είμαι σίγουρη. Πάλι λόγω ECR. Ελέγχουμε λοιπόν τη 15. Είστε οι ταραχοποιοί σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και σας ζητώ και συγγνώμη για αυτό που λέω. Λοιπόν, εγκρίνεται. Ωραία, πάμε στη 16 υπέρ. Κατά. Αποχές, το ίδιο πράγμα νομίζω εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 19. Υπέρ, κατά, Αποχές νομίζω εγκρίνεται. Τέλος. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά το σύνολο του σχέδιου νομοδότης. Άρχεται η ψηφοφορία. 14, let Exactly 14. 14, yeah. Um, simply that we vote anything which is not related to the common provision of regulation. And this year. And the final vote, and then we will vote in November. What do you mean? On this year. So, dear colleagues... Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε εδώ δεν έχουμε ψηφοφορία για όλα, γιατί υπάρχει συμφωνία να μην ψηφίσουμε τα recital 13, συμβαστική 2, στο άρθρο 5 επίσης συμβαστική 5 και στο άρθρο 11 συμβαστική 9. Το Νοέμβριο θα δούμε όταν έχουμε τη νέα τροποποιημένη εντολή. Στο CPR η λάβει ε, τον Ιούλιο, λέει η Πρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα ασυμβίβαστου με κάποιες τροπολογίες και θα δούμε τι γίνεται το Νοέμβριο, σε τι συμφωνία θα καταλήξουμε. Άρα Συμβαστικέ 2, 5 και 9 είναι οι μόνε που δεν ψηφίζονται. Όλα τα άλλα τα ψηφίζουμε. Μάρκο, παρακαλώ, μπορεί και εσύ να πει κάποια πράγματα. Συμφωνώ με τη διαδικασία ότι συγκεκριμένα άρθρα τα οποία τα αντιτίθεται σε αυτά τα που αποφασίσαμε στο Γενικό Κανονισμό, αυτά πράγματι να αναβληθούν. Όμως θα ήθελα παρακαλώ να γράψετε στα πρακτικά με απόλυτη σαφήνεια ότι όλες οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν επί του περιεχομένου σε ορισμένα σημεία. Και θα ήθελα σήμερα πραγματικά να το επαναλάβω αυτό, έτσι ώστε το Νοέμβρη να ψηφίσουμε για όλα αυτά, όπως ακριβώς ε, το συμφωνήσαμε. ο Λάμπερτ. Επίσης για τα πρακτικά, γιατί είναι πραγματικά σημαντικό αυτό που είπε τώρα ο Μάρκους, ότι δηλαδή συμφώνησε να μην ψηφίσουμε ας πούμε για το άρθρο 11. Εχθές ε, είχαμε πράγματι τις ε, επαφές με τους ε, άλλους εισηγητές και αποφασίσαμε να δεσμευτούμε για το περιεχόμενο. Αλλά είναι καλύτερα να ψηφίσουμε γιατί από τη μια ε, έχουμε την εντολή να μην ψηφίσουμε και από την άλλη λέμε θα ψηφίσουμε το Νοέμβρη. Άρα δηλαδή το θέμα είναι η νομική βάση που πρέπει να ισχύει. Δεν έχω διαφωνία επί του ουσίας, αλλά ε, να καταγραφεί ε, το τι θα γίνει, ε, να καταγραφεί στα πρακτικά το τι θα γίνει κατά την επόμενη ψηφοφορία. Ναι, αλλά δεν αρχίζουμε τώρα τη συζήτηση, Βίκτορ. Όχι βεβαίω συζήτηση. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επιβεβαιώσω ότι αν συμφωνήσουμε να αλλάξουμε την εντολή για τον κανονισμό Common Provisions και εγώ στην έκθεσή μου θα συμπεριλάβω ε, την ε, ίδια πρόταση για να υπάρχει συμβατότητα με τον κανονισμό αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία. 51 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 53 υπέρ, μισό λεπτό, 53 υπέρ κατά, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η, 4 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα δεν ψηφίζουμε για το άρθρο 5. Πάμε στη συμβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 Εγκρίθηκε η συμβαστική 6, άρα καταπίπτει. Πάμε στη συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 όχι η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 8 όχι, όχι όχι ψηφίζουμε ψηφίζουμε για την 8 τη συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 και 105 από κοινού. Όχι, πάμε στην 107 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το 11 φεύγει, δεν ψηφίζουμε γι' αυτό. Η 133, γι' 3 αυτήν ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 19 εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές, όχι με συγχωρείτε, 134, ελέγχουμε για την 134, ψηφίζουμε, απορρίφθηκε. Η 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές ε, νομίζω εγκρίθηκε. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά απορρι... αποχές απορρίπτεται, η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Εκτιμώντας 13 ε, δεν ψηφίζουμε. Πάμε στη 43 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία. Το Νοέμβρη δεν έχουμε τελική ψηφοφορία. Τελείωσαν οι ψηφοφορίες. Πω, πω. Άλλη μία ψηφοφορία έχουμε. Δεν μπορώ άλλο, λέει η πρόεδρος. Όλτζι Μπλάσακ. Όλτζι Μπλάσακ.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 αποχές. Νομίζω η ίδια κατάσταση ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Η 40 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω η ίδια κατάσταση, 41. Υπέρ, κατά, αποχές,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 αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατάποχες απορρίπτεται, η 7 υπέρ, κατάποχες εγκρίνεται, 49 υπέρ, κατάποχες εγκρίνεται, η 8 υπέρ, κατάποχες εγκρίνεται, η 50 υπέρ κατάποχες εγκρίνεται, 51 υπέρ κατάποχες εγκρίνεται, 52 υπέρ κατάποχες εγκρίνεται, 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά μισό λεπτό, μισό Ποιος είναι υπέρ της 9 παρακαλώ. Τώρα κατά, άρα εγκρίθηκε. Η 10 υπέρ κατά ε, απορρίπτεται αυτή. Η 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 15 υπέρ, μισό λεπτό, η 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 55 υπέρ κατάποχες απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά απορρίπτεται, 57 υπέρ κατά απορρίπτεται, 58 υπέρ κατά απορρίπτεται, 59 υπέρ κατά απορρίπτεται, 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκτιμώντας 18, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 21 υπέρ κατά ελέγχουμε για την 21. It's rejected 19 to 19. So we vote 22 in favor. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, οι δύο υπέρ, κατά, δεν ξέρω, νομίζω ότι απορρίφθηκε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. «24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 25 υπέρ κατάποχες εγκρίνεται, 26 υπέρ κατά εγκρίνεται, 27 υπέρ κατά εγκρίνεται, 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 3 υπέρ κατά απορρίπτεται, αλλά κάνουμε έλεγχο. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία. The vote is closed. No, not not. You repeat. You repeat. Sorry. No, it's okay. It's adopted. Yeah. You repeat again.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 Ladies and gentlemen, we should continue and the next item... Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι οι κοινέ διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και κατάρριση του κανονισμού 1083 του 2006 με συνεισηγητές την Κωνσταντσε Κρέλ και τον Λάμπρε Φανίστελ Ρόι. Κύριε Ματσόνη, θέλει τώρα το λόγο ή να δώσουμε πρώτο λόγο στους συζητητές μας και μετά σε σας κυρία Ματσόνη. Ναι, ξέρω τι πρόβλημα έχετε, κυρία Ματσόνη, αλλά να ακούσουμε πρώτα τους συζητητές. Λάμπερτ και μετά η Κωνσταντζ. Λάμπερτ, έχει το λόγο. Overall, uh, uh, Μισή ώρα έχουμε μόνο, να σας πω έτσι. Ε, γι' αυτό να είστε σύντομοι, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Πώς προχωράμε. Να σας πω, έχουμε την εντολή. Τη διατυπώσαμε τον Ιούλιο. Και αφού κάπως είχαμε μία συνάντηση για να δούμε προς τα που οδεύουμε, θα σας πω τώρα πώς έχει κατάσταση. Τι αποφασίσαμε. Έχουμε τριμερή διάλογο κάθε εβδομάδα. Πλην των Στρασβούργων. Από πλευράς μας λοιπόν έχουμε δώσει απόλυτη προτεραιότητα στο θέμα και χαίρομαι που έχουμε προχωρήσει. Βέβαια πρέπει να δούμε τις θέσεις μας ο ένας τον άλλον. Έχουμε και τη διαπραγματευτική ομάδα. Νίκο σκιώδη στο γενικό κανονισμό. Οι συγκητές αυτοί παρακολουθούν την κατάσταση. Έρχεται τα Και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε, όπως έχουμε αποφασίσει. Να κάνω ένα πιο γενικό σχόλιο. Ξεκινήσαμε με βάση την εντολή μας, αλλά πρέπει να σας πω ότι εν γέννη το Συμβούλιο δεν έχει καταλήξει για όλα τα στοιχεία της εντολής και πολύ σύντομα θα υπάρξει μια συνεδρίαση του Συμβουλίου και ελπίζουμε να σημειωθεί πρόοδος. Τα σημαντικότερα υποσυζήτηση θέματα αυτή τη στιγμή είναι η διατύπωση των άρθρων ορισμοί κτλ. Έχουμε μιλήσει για την αρχή της εταιρικής σχέσης και τώρα ξεκινάμε το κομμάτι προγραμματισμού. Μέχρι στιγμής, ίσως θα περίμενε κανείς να έχει συμμεθεί μεγαλύτερη ναι. πρόοδος, για να μην στο λεφτό, αλλά νομίζω ότι εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε τη μετάφραση των άρθρων που δεν ψηφίσαμε τον Ιούλιο, για το Γενικό Κανονισμό συγκεκριμένα και να προετοιμάσουμε τώρα την ψηφοφορία για τις ετολογικές σκέψεις, τα recitals. Έτσι έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή. Όχι και πολύ πρόοδος. Παρ' όλα αυτά έχουμε τουλάχιστον συζητήσει πολλά άρθρα για να δούμε αν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση του το Συμβούλιο. Εμείς από τη δική μας θέση, τις βασικές μας αρχές δεν έχουμε μετακινηθεί καθόλου αυτή τη στιγμή. αυτό ω γενική εισαγωγή. Η Κωνσταντζε ενδεχομένως να έχει να προσθέσει κάτι περισσότερο. Όχι πολλά, σύντομα. Η αρχή της εταιρικής σχέση θα είναι από τα πιο δύσκολα που θα χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Βασικά συμφωνούν και αυτοί, αλλά θα γίνουν τα πράγματα όλο και πιο δύσκολα γιατί δεν προτείνουν τίποτα. Η Κομισιόν έκανε πρόταση, εμείς είπαμε να το ελέγξουμε, να το συζητήσουμε, είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση, αλλά δεν έγινε τίποτα, δεν το συζητούν. Λίγη πρόοδος λοιπόν, αλλά όχι όσοι θα θέλαμε. Σας κατευχαριστώ για τις πληροφορίες αυτές. Η κυρία Ματσόνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ζήτησα το λόγο να μιλήσω γιατί πρόκειται για μια... Ε, παρέμβαση που είναι περισσότερο θέμα μεθόδου και όχι τόσο επί της Θέλω λοιπόν να στηρίξω τους ε, συντάκτες αυτής της έκθεσης αλλά και άλλων κανονισμών γιατί θεωρώ ότι η τριμερή συνάντηση θα πρέπει να φτάσει στη θέση με την οποία είχε ξεκινήσει από την αρχή. Δηλαδή να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ε, της τριμερούς όλοι οι συγητές και με κανονισμών και ε, να μοιράζεται ο χρόνος με ανάλογα με θεματικές ενότητες και όχι με κανονισμούς. Για την 2014-2020, ε, για αυτή την περίοδο, ε, θα μπορούσε να υπάρξει ένας γενικός κανονισμός, ο οποίος ε, θα αναδιατυπώνει όλα τα βασικά σημεία και μετά διάφοροι υποκανονισμοί. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συμμετοχή τόσο για να εξετάσουμε τις, ε, τα διάφορα σημεία όσο και για να επιταχύνουμε την ε, διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή εγώ εδώ έχω επέμβει επανειλημμένα για αυτό το επιχείρημα και η, το Προεδρείο μου είχε πει ότι θα προχωρούσαμε όπως είχε συμφωνηθεί στην αρχή της συμφωνίας, δηλαδή ένα θεματικές ενότητες και όχι ανακανονισμό, θέλω να ρωτήσω την αρχή τι συνέβη, μήπως είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί η στάση σας. Και εγώ θέλω να πω ότι συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος. Να δούμε δηλαδή κατά πόσον σε θέματα μεθόδου είναι δυνατόν να ε, προχωρήσουμε ανά θεματικές ενότητες. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χρήσιμο για μια συζήτηση η οποία θα μπορούσε να ε, ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Η κυρία Κρέλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Μάρκους. Πράγματι υπήρξε κάποια συζήτηση και υπήρξε και μία προκαταστική ε, συνεδρίωση αμέσως μετά την 11η ε, ή την 12η Ιουλίου, δεν θυμάμαι πια. Και τελικά ε, συμφωνήσαμε ότι θα προχωρήσουμε με θεματικές ενότητες. Θα ξεκινήσουμε με τις πρώτες αυτές ενότητες και μετά θα ακολουθήσουν οι άλλες ε, διαπραγματευτικές ομάδες. Η Ντανούτα Χούπνερ τα ανέφερε αυτά. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Όταν υπάρχει ανάγκη σε ορισμένα θέματα, θα πρέπει οι συνάδελφοι από άλλες ε, ομάδες να προσκαλούνται και αυτοί. Αυτό ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε και εντωμεταξύ έχουμε φτάσει στο δεύτερη, στη δεύτερη τριμερή. Νομίζω ότι και οι άλλοι προετοιμάζονται ε, σιγά σιγά, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι σιγά σιγά προτιμάμε τις ε, θεματικές ενότητες. Um, Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να προχωρήσουμε σε όλα τα επίπεδα. Όπως στην καλύτερη δυνατή παλιροφόρηση. Η Κωνσταντσα ήδη είπε ότι θέλουμε επιτάχυνση και να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τα, τους διαφορετικούς κανονισμούς. Από ό,τι ξέρω, ήδη υπάρχουν σχέδια προγραμμάτων για τις διαπραγματεύσεις. Δεν είναι αλήθεια λοιπόν ότι τίποτα δεν γίνεται. Υπάρχει σαφή σχέση μεταξύ του γενικού κανονισμού και των υποκανονισμών του. Προς Ίσως υπάρχει η παρεξήγηση ότι τα παίρνουμε όλα μαζί, ενώ όχι, υπάρχουν διαφορετικές διαπραγματευτικές ομάδες. Είμαστε ανοιχτοί για πληροφόρηση, ίσως μπορούμε να το αναφέρουμε αυτό και στον πρόεδρο. Να ζητήσουμε αν μπορούν να έρθουν να ακούσουν και άλλοι εισηγητές ας πούμε. στοχεύουμε τον Νοέμβριο Ίσως καλό θα ήταν να μας πει και η Κομισιόν να επαληθεύσει αν ο δημοσιονομικός κανονισμός μπορεί να γίνει και αυτός αντικείμενο κάποιας πληροφόρησης. για το δημοσιονομικό κανονισμό. Ίσως ένα-ένα να πρέπει να τα βάλουμε στο δικό μας κείμενο, δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτω και ίσως η Κομισιόν να μας το λύσει. Μισό λεπτό. Ε, θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Ματσόνη να μας πει κατά πόσον οι απαντήσεις που δόθηκαν, κατά πόσον είναι καλές αυτές οι απαντήσεις ή μήπως εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα. Ε, γιατί και εγώ θυμάμαι ότι αυτό το θέμα των ε, θεματικών ενωτήτων ε, θέλαμε να το συζητήσουμε, να παρίστανται κάθε φορά οι συγητές. και από τη δική μου την πολιτική ομάδα μου είπαν ότι αυτό δεν λειτουργεί όσο και αν σας εκνευρίζει, να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Έτσι κι αλλιώς εδώ πολλά γίνονται χωρίς διαφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν ας μην προσθέτουμε άλλο ένα. Θα ήθελα τώρα η κυρία Ματσόνη να τοποθετηθεί πάνω σε αυτές τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είμαι ικανοποιημένη. Επί της ουσίας δεν συμφωνώ. Γιατί όπως ήδη σας είπα, θα προτιμούσα να κάνω αυτό που είχαμε πει στην αρχή. Δηλαδή, στις διαπραγματεύσεις να συμμετέχουν όλοι εκείνοι που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν. Βέβαια, ίσως και σε αυτήν την περίπτωση, επειδή ίσως ψηφίστηκε ένα συμβασμός ε, λανθασμένα, να υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Εγώ προσωπικά παρενέβην δύο φορές όταν συζητάγαμε ε, για οργανωτικά θέματα. Αυτό συνέβη τελευταία φορά τον Ιούλιο. Θα έπρεπε να κάνουμε αυτό που είχαμε πει στην αρχή, να ε, προχωρήσουμε με θεματικές ενότητες και όχι με κανονισμούς. Ε, από ό,τι φαίνεται, η κυρία Κρέλη κάτι άλλο, μάλλον υπάρχει εδώ πρόβλημα συνεννόησης. Εγώ επιμένω στέση Πρέπει να φύγω σε ένα λεπτό, αλλά μία σύντομη πληροφόρηση. Η διαπραγματευτική ομάδα για το ERDF δεν έχει ακόμα τις τελικές ημερομηνίες. Δεν τις έχει επιβεβαιώσει το Συμβούλιο και η Επιταροπή. Έπειτα έχω την πληροφορία από, το, από την κυρία Χιούμπνερ ότι οι εργασίες για το CPR θα οργανωθούν ως εξής. Οι κύριοι εισηγητές και εισηγήτριες βήμα το βήμα θα καλέσουν τους εισηγητές και εισηγήτριες για τους τομεακούς κανονισμούς για να συνεννοηθούν. Αυτά μου έφτα εγώ. Και περιμένω και εγώ ως εισηγητής για το Περιφερειακό Ταμείο να μάθω τις ημερομηνίες που αφορούν το Περιφερειακό Ταμείο. Από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει η ιδέα να κληθούν όλοι οι συγητές σε όλες τις συνεδριάσεις, αλλά να κληθούμε εμείς οι συγητές για τα συγκεκριμένα θέματα όποτε εμφανιστούν. Αυτό έμαθα εγώ. Και περιμένω να μάθω σε ποια συνεδρίαση θα κληθώ. η Κοιτάξτε, αυτή είναι η συμφωνία ότι οποτεδήποτε προκύπτουν θέματα τα οποία αφορούν άλλους κανονισμούς, εκεί να ε, προσκαλούνται και οι συγητές. Πράγματι αυτή είναι η συμφωνία. Το πρόβλημα που τίθεται όμως είναι ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο βασικό θέμα. Και αυτό είναι αρμοδιότητα που έχει, είναι θέμα που έχει σχέση με τον βασικό κανονισμό. Και παρότι λοιπόν παρακαλέσαμε το Συμβούλιο να μας δώσει κείμενο, ε, νομίζω ότι δεν έχουμε καταλήξει ούτε καν σε αυτό. Δηλαδή ε, δεν μπορούμε να ε, κάνουμε περισσότερα από αυτά που είπε προηγουμένως ο Λάμπερτ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν προσφέρθηκε η δυνατότητα να, έχουμε, να προσκαλέσουμε τους ηγητές από κάποιον άλλο κανονισμό. Γι' αυτό λοιπόν πράγματι ε, συμμερίζομαι τις ανησυχίες του Λάμπερτ ότι η όλη διαδικασία ε, καρκινοβατεί. Αν συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με τον τρόπο αυτό, αυτό δεν οφείλεται σε εμά. Σε μας ε, έχουμε πει στο Συμβούλιο ότι ε, ε, το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο η αν θέλετε Προεδρία είναι εκείνη που σε πολύ απλά θέματα λένε ότι μισό λεπτό να δω τώρα αν η ομάδα του Συμβουλίου ε, θα μου δώσει εντολή ή όχι. Το όλο θέμα είναι πολύ άκαμπτο. Ε, προφανώς στα εξειδικευμένα θέματα οι συνάδελφοι είναι προσκεκλημένοι. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε ε, αυτήν την πληροφορία και θα ήθελα μεταξύ σας ε, κάπως να τα βρείτε Να δούμε λοιπόν μήπως μπορεί να γίνει κάτι. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν θα δώσω το λόγο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια σύντομη πληροφορία η διαπραγματευτική ομάδα για τον κανονισμό για τη συνοχή ακριβώς στην διακατάσταση βρισκόμαστε. Έχουμε προτείνει διάφορες ε, ημερομηνίες για τις ε, τριμερείς μας συναντήσεις, αλλά δεν έχουμε από πλευρά Συμβουλίου καμία απάντηση ακόμα. Και όταν έχουμε θα, σκηνε, θα έχουμε πλέον την ημερομηνία για να ξέρουμε πότε θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις και θα δούμε μετά πώς μπορούμε το πρόγραμμα με το, για τις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό της κοινή διατάξης να το εντάξουμε στο πρόγραμμα. Κύριε Μπέρκοβιτς, σας βλέπω εδώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, θα είμαι σύντομος. Είναι λίγο τεχνικό το θέμα και ίσως να γίνει πολύπλοκο και ζητώ την κατανόησή σας και την υπομονή σας, αλλά να πω κάτι για το CSF, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Έχουμε μια τροποποιημένη πρόταση για τον κανονισμό για να λάβουμε υπόψη τη απόψεις του Κοινοβουλίου και θέλουμε βέβαια να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο για την ολοκλήρωση του θέματος. Έχουμε ένα παράρτημα και προτείνουμε και κατεξουσιοδότηση πράξη που ουσιαστικά θα περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά στοιχεία. Τώρα, έρχομαι στο ζήτημα της προσαρμογής. Λόγω της συμφωνίας για τον αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό, πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί το κείμενο. Και πρέπει να θυμίσω την αφετηρία. Ποια ήταν η αφετηρία της Κομισιόν και για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και για τον κανονισμό ε, των κοινών διατάξεων. Ήταν ε, οι συστάσεις ε, στην απαλλαγή του 2010 όπου ζήτησε το Κοινοβούλιο να κάνουμε ως Επιτροπή ό,τι μπορούμε λόγω και των νομοθετικών πλαισίων που δεν δίνουν στα κράτη-μέλη κίνητρα για να συμμορφωθούν προς τους κανόνες, ούτε και η Κομισιόν έχει τα απαραίτητα εργαλεία στη διάθεσή της για να ε, επιβάλλει μάλιστα και καιρό σε περίπτωση με συμμόρφωση. Ζήτησε λοιπόν το Κοινοβούλιο από την Επιτροπή να ενισχύσει τον αποπτικό τη ρόλο και να δημιουργήσει αποτελεσματικού μηχανισμού επιβολή κυρώσεων ώστε να μπορεί να αναλάβει και να φέρει σε πέρα στην ευθύνη τη για την υλοποίηση του προπολογισμού. Οι συστάσει επίση περιλάμβαναν και ορισμένε συγκεκριμένε προτάσει μεταξύ αυτών την εφαρμογή καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων. Αυτά προσπαθούμε να κάνουμε με τις προτάσεις μας. Σε ό,τι αφορά τώρα την αρχιτεκτονική για τη διαχείριση τη δημοσιονομική και τον δημοσιονομικό έλεγχο, τα βλέπετε αυτά τα στοιχεία. Πρώτον, μια σταθερή βάση για τη διασφάλιση, τη βεβαίωση που δίνει η Επιτροπή, το assurance και έχουμε ένα σύστημα λογαριασμών ε, που εξετάζεται και γίνεται ή δεν γίνεται αποδεκτό για να έχουμε την απαραίτητη διαβεβαίωση για τη μετήσια έκθεση πρόοδου ε, της Κομισιόν, ένα σύστημα αποζημίωσης που κρατάει το 10% μέχρι να ολοκληρωθεί ο εθνικός κύκλος ελέγχου και αυτό αντισταθμίζεται με μια προχρηματοδότηση για να έχουν την απαραίτητη ταμιακή ροή και έπειτα υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών να ε, αποζημιώσουν τους δικαιούχους πριν δηλώσουν τις δαπάνες τους στην Κομισιόν. Κίνητρο για να έχουν τους έγκυρους έλεγχους. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον ενισχυμένο οπτικό ρόλο της Κομισιόν, έχουμε την εφαρμογή πλέον συστηματικών διατάξεων διορθώσεων μετά ε, την ανείχνευση σφαλμάτων, είτε από την Κομισιόν είτε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν θέλουμε να επιστρέφουν περισσότερα χρήματα με αυτόν τον τρόπο, αλλά να δημιουργήσουμε κίνητρα ώστε τα κράτη-μέλη να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Υπάρχει μια αλλαγή επίση που προτείνουμε σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνονται τα συστήματα σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει μια πρόταση να υπάρξει ένα σύστημα, θέλετε, διαπίστευσης, δηλαδή βάσει ευρωπαϊκών κριτηρίων. Ποια είναι η σημαντική αλλαγή που προτείνουμε εδώ. Αρμόδιο το, κράτο, το κράτος μέλος και το η Επιτροπή παίρνει μία προσέγγιση εδραζόμενη στους κινδύνους. Risk-based. Ναι. Κατά την άποψή μα, εμεί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε του πόρου μα και τα μέσα μα για να στοχεύσουμε εκεί που υπάρχουν οι υψηλότεροι κίνδυνοι, αυτού του τομεί. Και βέβαια όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και εύκολα το να εντοπίσει κανεί του πιο προβληματικού τομεί. Λοιπόν, κατ' ουσίαν αυτά είναι επιτάπητο. Δεν έχουν αλλάξει τα περισσότερα από αυτά. Σίγουρα στόχο τη Κομισιόν είναι να μην αλλάξει και δεν έχουν αλλάξει οι στόχοι του, του κοινού στρατηγικού πλαίσιου. Μετά τι αλλαγέ βέβαια στον δημοσιονομικό οργανισμό έχουν γίνει κάποιε αλλαγέ και εδώ, αλλά εν συντομία θα σα πω τα σχετικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέταση και την αποδοχή, την έκδοση των λογαριασμών, χρειάζεται να γίνουν αλλαγέ. Πρώτα απ' όλα, ο δημοσιονομικό κανονισμό δεν μιλά πια για καθάριση των λογαριασμών, clearance. Πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε τη διαδικασία, να έχουμε την έγκριση των λογαριασμών. Απλή λογιστική διαδικασία αποσυνδεδεμένη από θέματα νομιμότητα και κανονικότητα. Επίση, πρέπει να διευκρινίσουμε τι διαδικασίε. Ωστόσο, δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν πολλέ πτυχέ του συστήματο, μεταξύ αυτών το σύστημα δημοσιονομική διαχείριση, η διακράτηση αυτή το 10% του στου δικαιούχου κτλ. Έρχομαι στον ορισμό των αρχών που θα είναι αρμόδιες για τη διαχείριση και τον έλεγχο. Η πρώτη αλλαγή που θα πρέπει να λάβει η χώρα είναι ότι ο όρος accreditation πρέπει να αντικαταστεί από τον όρο designation, όχι διαπίστευση αλλά ορισμός. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τώρα που ε, δημιουργούν άλλη επικαλύψεις στο δημοσιονομικό κανονισμό. Μπορούμε να τα διαγράψουμε και αυτά. Επίσης πρέπει να δούμε κατά πόσον υπάρχει ανάγκη δοκιμαστικής περίοδου ή όχι. Πάντως, αυτό που δεν χρειάζεται να αλλάξει είναι η διαδικασία ορισμού των αρχών ε, διαχείρισης πιστοποίησης με βάση τη γνωμοδότηση ανεξάρτητης ε, αρχής ελέγχου, ούτε τα κριτήρια για τον ορισμό πρέπει να αλλάξουν. Όπως σας είπα και πριν, δεν υπάρχει ανάγκη, κατά την άποψή μας τουλάχιστον, να αλλάξει η διαδικασία που είχαμε προτείνει για την εκτίμηση, την αξιολόγηση της διαδικασία αυτής ορισμού από την Κομισιόν. Για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημα του κ. Φανίστελ Ρόι. Κατά την άποψή μας, σχετικά είναι τεχνικό το εγχείρημα, πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές, δεν είναι όμως ε, κάτι που θα αλλάξει το κείμενο και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα. Ευχαριστώ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να τα επεξεργαστούμε σε αυτή τη βάση. Μετά και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια και θα δώσουμε το κείμενο που μπορεί να συζητηθεί και να ψηφιστεί. Άρα το χρονοδιάγραμμά μας δεν αλλάξει περαιτέρω. Αν υπάρξουν τίποτε απρόβλεπτα θα το δούμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την Επιτροπή και τον εισηγητή μας ε, για την ενημέρωση. Και πάμε τώρα στην έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Λίγης, υλοποίηση και εφαρμογή. Η κυρία ε, Φεραγκούτ ε, θα μας ενημερώσει για την έκθεση αυτή. Κοιτάξτε, στη Βαλένθια, καθώς και στη Γαλλικία και τη Μούρθια, έγιναν και ηλικές και ανθρώπινες ζημιές σημειώθηκαν και ιδιαίτερα στη Λόκα και Φουέρτα Λουμπρέρα, στη Μουρθία. Η Μούρθια. Υπήρξαν μαζικές απώλειες, ζωές, σχολεία, αγροκτήματα, άλλα κτίρια, βιομηχανίες, μαγαζιά και θα ήθελα να αρχίσω την παρέμβαση μου αυτή για το Ταμείο Αλληλεγγύης αναφέροντας τα θύματα και την υποστήριξη για τις οικογένειές τους. Το πρόγραμμα υπάρχει εδώ και 10 χρόνια από το 2002 και νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό, πολύ καλό εργαλείο, όλοι το είπαν αυτό. και 49 περιπτώσεις επίγουσας βοήθειας χορηγήθηκαν μέσω εκείνου. Πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν, αν θα θυμάστε καλά, για το σεισμό στην Ακουήλα στην Ιταλία και ήταν το υψηλότερο ποσό που πληρώθηκε ποτέ για τέτοιο σκοπό. Το Ταμείο Αλληλεγγύης όμως, τα τελευταία 10 χρόνια, είχε και ορισμένα προβλήματα. Εύρος, πεδίο εφαρμογής κτλ. Γι' αυτό έγινε και η αναθεώρηση το 2005 η Κομισιόν πρότεινε την αλλαγή της λειτουργίας του Ταμείου και συμφώνησε και το Κοινοβούλιο. Τελικά όμως η Κομισιόν αναγκάστηκε να αποσύρει την ομοθετική της πρόταση. Τώρα είμαστε σε θέση να προτείνουμε βελτιώσεις στη λειτουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης, ιδιαίτερα μετά από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2008 που ανέφεραν και αυτοί τις θεομηνίες και είπαν ότι είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί κανείς στις ελπίδες που είχαν δημιουργηθεί στις προσδοκίες. Και όλοι επέκριναν το γεγονός ότι το εργαλείο αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί πολύ γρήγορα και γι' αυτό πρόσφατα η Κομισιόν άρχισε να κάνει μία νέα αναθεώρηση και τον Οκτώβριο του 2011 αποφάσισε να πάρει μερικά μέτρα για να μειωθούν οι ελλείψεις στη λειτουργία του προγράμματος και να λυθούν μερικά προβλήματα. Δεν σκοπεύει όμως να αλλάξει τα ποσά που διατίθενται. Γι' αυτό έγραψα και εγώ την έκθεσή μου που αναφέρει αυτά τα 10 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας του Ταμείου που έχει επιδείξει αλληλεγγύη με όλους τους πληθυσμούς και περιφέρειες που έχουν πληγεί από θεομηνίες και είχε και πολύ θετική αξιολόγηση από την κοινή γνώμη. Επίσης τονίζω ότι έχει φανεί, έχουν σημειωθεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις πολλές φορές και ότι είναι δύσκολο να πρέπει να συμφωνήσουν και οι Κομισιόν και το Κοινοβούλιο γιατί αυτό καθυστερεί τα πράγματα στην ανάλυση. Πολλές φορές οι πληρωμές γίνονται 9 ή 10 μήνες μετά την καταστροφή και άλλους δύο μήνες για να υποβάλει το κράτος την αίτηση κλπ. και ο ορισμός που χρησιμοποιώ είναι ότι πρόκειται για καταστροφές που δεν οφείλονται στην ανθρώπινη παρέμβαση γιατί εκεί θα υπήρχαν ασφαλίσεις. 70% των ετοιμάτων που υποβλήθηκαν ήταν αφορούσαν φυσικές καταστροφές στις περιφέρειες αλλά μεν αλλά απορρίφθηκαν γιατί ο κανονισμός είναι ασαφής ως προς το τι είναι μια περιφερειακή καταστροφή ή θεομηνία. Γι' αυτό ζητώ αποσαφήνισή του. Να, είμαστε, να, ξέρουμε τι λέμε όταν μιλάμε για περιφέρεια που έχει υποστεί φυσική καταστροφή, παραδείγματος χάρη σοβαρή περίπτωση ξηρασίας, καταστροφές που εκτιλήσονται μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα ο προηγούμενος ορισμός ήταν 10 εβδομάδες από την εμφάνιση του αρχικού προβλήματος. Αν διατηρείται θεωρείται φυσική καταστροφή. Αλλά για φαινόμενα όπως η ξηρασία χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να σημειωθεί, για να διαπιστωθεί το φαινόμενο. Τώρα όλα αυτά πρέπει να γίνουν βέβαια χωρίς να πειράξουμε τα ποσά, να μείνουν τα ίδια στον προϋπολογισμό. Ζητάμε πάντως να μειωθούν τουλάχιστον ε, να αυξηθεί η ταχύτητα αντίδρασης του Ταμείου, να μειωθεί η γραφειοκαρατία και να δίνονται ταχύτερα οι πληρωμές και τα, να λαμβάνονται τα υπόλοιπα μέτρα ταχύτερα. Προηγουμένως η διαδικασία ήταν πάρα πολύ αργή και μακρόσυρτη μέχρι να αποφασίσει κανείς την πληρωμή και μετά ακόμα παραπάνω για να γίνει η πληρωμή. Τώρα προβλέπονται ορισμένες προκαταβολές πάνω στην αίτηση για βοήθεια γιατί πολλές φορές οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές αντιμετωπίζουν επίσης πολύ δύσκολες καταστάσεις και γι' αυτό είναι βασικό οι πληρωμές να γίνονται γρήγορα, ίσως με προκαταβολές. Ο ορισμός της φυσικής καταστροφής, ξαναείπα, πρέπει να ξεκαθαριστεί και να καθοριστούν ακόμη σαφέστερα και οι πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του. Για να υπάρξουν σαφή κριτήρια η Κομισιόν καθόρισε το 1,5% του περιφερειακού ΑΕΠ στο επίπεδο ΝΑΤΣ 2 Είχαμε συγκρίνει το, την ανάγκη να υπάρχουν σαφή κριτήρια, αλλά αυτό το ποσοστό είναι λίγο ψηλό. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος αν μπορεί να προσφύγει στο ταμείο. Και γι' αυτό εμείς προτείνουμε το ποσοστό αυτό να είναι χαμηλότερο. Νομίζω γενικά ότι ό,τι έχει να προσφέρει κάθε πολιτική ομάδα ως πρώτα θα εμπλουτίσει το γενικό κείμενο. Υπάρχει πρόβλημα βέβαια, επειδή έχουμε την οικονομική κρίση. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα και να επιταχύνουμε την κατάσταση. Και θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το Ταμείο θα έχει πραγματικά πολλά να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ για την επισκόπηση αυτή την ενδιαφέρει. Θέλει, θέλει κάτι να πει κανεί, κάτι. Κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα, το συζη... θα το συζητήσουμε, θα το πάμε το θέμα αυτό το οποίο αναβλήθηκε κάπου αλλού. Πρόεδρος. Το μόνο που μου είπαν είναι να δώσουμε προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών και να μην συζητηθεί το θέμα σας τώρα. Συμφωνείτε, μάλιστα. Κωνσταντσε, για την έκθεση αυτή που συζητάμε τώρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Σταυρακάκης δεν μπορούσε να είναι εδώ και όδηση εισηγητής για το Ταμείο Λεγγύης και μου ζήτησε να δώσω την απάντησή του σε εσάς. Πρώτα απ' όλα, κ. Σταυρακάκης θέλει να ευχαριστήσει για την ε, πολύ καλή έκθεση της στην εισηγήτρια. Το Ταμείο Αλληλεγγύης θεωρεί ότι είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα εργαλεία αλληλεγγύης που έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προστιθέμενη αξία αυτού του Ταμείου βέβαια είναι πολύ μεγάλη, ιδίω από τη στιγμή που χρειάζονται προσπάθειε λιτότητα αυτή τη στιγμή, δημοσιονομική προσαρμογή από τι περισσότερε χώρε. Στην έκθεσή της ε, η συγκεκριά προτείνει τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό της έννοιας των φυσικών καταστροφών. Πρέπει επίσης να θεσπιστούν γενικά κριτήρια για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των ε, ζημιών. Αναγνωρίζεται η δυσκολία ε, του να έχουμε έναν ενίο ορισμό για τις καταστροφές, παρόλα αυτό αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε καλύτερα δυνατόν τις επιλέξιμες καταστροφές και έτσι θα μειώσουμε και τον αριθμό των ε, αιτήσεων που λόγω μη επιλεξιμότητας απορρίπτονται. Θέλει επίσης να τονίσω ότι υποστηρίζει τη θέση της εισηγητρίας ότι το Ταμείο θα πρέπει να συνεχίσει όταν υπάρχουν ε, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να παρεμβαίνουν ακόμη και αν δεν φτάνει η καταστροφή αυτή το κατόφλι της επιλεξιμότητας. Πρόσφατα ε, ξέρουμε ότι κινητοποιήθηκε πολλές φορές το Ταμείο για να παράσχει βοήθεια σε πληγέντες υποψίες καταστροφές στα κράτη-μέλη, αλλά η διαδικασία ενεργοποίησης ε, και κινητοποίηση του Ταμείου είναι χρονοβόρα όπως αποδείχθηκε. Και έτσι δεν φτάνουν σε έφθετο χρόνο οι πόροι στους πληγέντες. Επομένως πρέπει να βελτιωθεί και η αποτελεσματικότητα αλλά και η ευελιξία του Ταμείου με απλούστευση των κανόνων και δικασιών που το διέπουν. Έτσι θα μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από την καταστροφή μέχρι τη χωρίς βοήθεια. Ας μην ξεχνάμε ότι η ταχύτητα της κινητοποίησης αυτού του Ταμείου αλληλεγγύη, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο βέβαια θεωρεί ότι δεν υπάρχει έγκαιρη παρέμβαση αυτού του ταμείου. Είναι πολύ καλέ οι προτάσει τη ηγήτρε επίση ό,τι αφορά την αύξηση τη ευελιξία του ταμείου που μπορεί να μα βοηθήσει να βρούμε λύσει για να μπορεί το ταμείο να βοηθήσει πιο αποτελεσματικά του πληγέντε. Τέλο, Θέλω να εκφράσω την συμφωνία μου με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Ταμείο να μείνει εκτός του δημοσιομικου πλαισιου πλαισίου 2014-2020 διότι πρέπει να ανταποκρίνεται και σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Άρα πρέπει να εξασφαλίσετε παρκή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Well done, Σε ευχαριστώ, Κωνσταντσε. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ. Η συγκίτρια έχει κάποιες παρατηρήσεις. Να δευτερολογήσει την κυρία Φέραγκουτ. Ευχαριστώ. Όχι, το μόνο που θέλω να ευχαριστήσω την Κωνστάνθα και περιμένω τις τροπολογίες όλων σας για να προχωρήσω στη σύνταξη της νομοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω κάτι θέλει να πει και η Κομισιόν, λέει ο Πρόεδρος. Όχι. Α, όχι. Ωραία. Τότε να πούμε την προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών για αυτήν την έκθεση 17 Οκτωβρίου για τις τρεις εκθέσεις τώρα που δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Πρέπει να πούμε όμως ποιες είναι οι προθεσμοί της κατάστασης τροπολογιών. Σε ό,τι αφορά την έκθεση της κυρίας Ρούλε, προθεσμία 27 Νοεμβρίου. Έκθεση Μάνκα, πάλι το ίδιο, 27 Νοεμβρίου. Και Λένα Κολάρας Καμπομπίνσκα, 26 Νοεμβρίου του τρέχοντος. Η προθεσμία σας, κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Απλά για όσους έχουν απομείνει τους ολίγους, να πω ότι αύριο έχουμε μια συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια, να σας το επενθυμίσω και να κηρύξω την λήξη της σημερινής συνεδρίασης.